Λοιπόν, να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε αντίρρηση. Um, λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι η παρουσίαση από τον Γενικό Διευθυντή Ματίας Ρούτε για την ε, Ομάδα Δράσης Μεσογείου, Task Force Mediterranean. Είναι μία ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα. Όπως βλέπετε είχαμε μία Ιταλική παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ιταλικής ε, Προεδρίας. Αλλά η ουσία της σημερινής ημέρας είναι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Και είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω τόσες πολλές παρουσίες. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τις ελληνές διακοπές και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ και ε, Ελπίζω να έχουμε και θα έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας να μιλήσετε, ιδίως εκείνοι όσοι δεν μπόρεσαν να μιλήσουν στην τελευταία ε, συνεδρίαση. Εισαγωγικά ήθελα να πω ότι αυτή η ομάδα δράσης ε, Μεσογείου ε, δημιουργήθηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων στις 7-8 Οκτωβρίου του περασμένου έτους για το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Λαπεντούσα στις 3 Οκτωβρίου 2013 και υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας της Κομισιόν για την υλοποίηση αυτής της ανακοίνωσης, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί κατά διάφορους τρόπους και αυτή τη στιγμή και ε, έχει συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής και ε, ο εισηγητής ε, Ματία Ρούτε, ο οποίος ε, είχε εργαστεί παλαιότερα και στη Γενική Διεύθυνση ενέργεια, τώρα είναι επικεφαλής της γενική διεύθυνση στην Κομισιόν Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα μα ενημερώσει βέβαια η Τελική Προεδρία έχει την ευθύνη ε, και είναι επικεφαλής τη όλη προσπάθεια και θα ήθελα και εγώ να παρέμβω πριν δώσω το λόγο στα μέλη μας. Οπότε λοιπόν δίνω το λόγο με τη σειρά. Καταρχάς τον κύριο Ρίτε ε, για να μας μιλήσει για αυτή την ε, ομάδα δράσης. Εν συνεχεία στην Ιταλική Προεδρία, εν συνεχεία θα μιλήσω και εγώ, μετά θα μιλήσουν τα μέλη. είπα το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριο Ρούτε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και καλό σα απόγευμα, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ καταχάς που με καλέσατε για την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και σε εσά, Πρόεδρε, για την εκλογή σας. Όπως είπατε ήδη, ε, είμαι το καινούριο παιδί στη γειτονιά. Ε, δύο μήνες έχω αναλάβει αυτή τη θέση στο, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Βεβαίως ενημερώνουμε ε, εις βάθος. Έχω μάθει ήδη πάρα πολλά, δεν ξέρω αν τα έχω μάθει όλα, οπωσδήποτε όχι όλα, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσετε, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο του διορισμού μου. Θα αναφερθώ σε ορισμένα ουσιώδη θέματα και συνεχεία θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας μέσα στα πλαίσια της συζήτησης και να μάθω κιόλα να ενημερωθώ από τις ερωτήσεις σας για να κατανοήσω περισσότερο τις απόψεις σας. Συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα ε, της, ε, των μεταναστών είναι το βασικό θέμα που θα απασχολήσει την θητή αυτή του Κοινοβουλίου και του ε, ε, Προέδρου του Σώματος ε, και ακριβώς αυτό το δείχνει και η παρουσία μου εδώ για να ενημερώσω για το έγγραφο εργασίας που συνέταξε τα στελέχη μου για την ομάδα δράσης Μεσογείου και ε, ε, σκέφτομαι αυτές τις μεταναστευτικές ροές ε, τους τελευταίους μήνες και ιδίω αν κοιτάξετε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Δυτική Μεσόγειο. Αν δείτε στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου τι γίνεται με, τις με την αστασή κατάσταση που υπάρχουν εκεί, το πρόβλημα θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο πρόεδρος σας ενημέρωσε σύντομα όσον αφορά ε, το, ιστορικό της ομάδας δράσης ε, και δεν θα σας κουράσω ε, διαβάζοντας τις 44 σελίδες ε, του εγγράφου εργασίας ή τις πάνω από 200 δράσεις που περιλαμβάνει το ίδιο έγγραφο. Δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω, αλλά σας διαβεβαιώ ότι περιλαμβάνει, αναφέρει πάρα πολλές συγκεκριμένε δράσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, στο επίπεδο ε, ε, Υπουργών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να θέσουμε οπωσδήποτε ορισμένες προτεραιότητες. Προτεραιότητες σχετικά με τις δράσεις που θα πρέπει να, ανα, αναλυφθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και ο καλύτερος τρόπος για να ομαδοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες είναι τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που θα πρέπει να καλύπτουν τις τρίτες χώρες. Πρώτος πυλώνες λοιπόν τρίτες χώρες από, και θα περιλαμβάνουν τα περιφερειακά προγράμματα, ε, κινητικότητα, ε, λαθρέα διακίνηση ατόμων, ε, λαθρό μετανάστευση, μετανάστευση και το πώς θα επικοινωνούμε για να αξιολογούμε τα... και να αναλύουμε τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα του, μετα... μεταναστευτικού θέματος γενικά. Ο δεύτερος πυλώνας θα καλύπτει θέματα με τον έλεγχο των συνόρων και με το μεσογειακό με την μεταμεσογειακή κατάσταση αν θέλετε, το post mare nostrum. Πέρσι τον Οκτώβριο είχαμε αυτή την ε, φοβερή τραγωδία στη Λαπεντούσα με πάνω από 360 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος που πνίγηκαν και τους πρώτους μήνες αυτού του έτους είχαμε πάλι εκατοντάδες σήματα σε, από ανθρώπους που πνίγηκαν προσπαθώντας με 160 160 είναι οι καταγεγραμμένοι, ε, τα καταγεγραμμένα θύματα. Οι άνθρωποι δηλαδή που πνίγηκαν όταν προσπαθούσαν το διάφορων σκαφών να περάσουν ε, απέναντι και να διανύσουν αυτή τη θάλασσα που τη δική μας, το Μάρε Αυτή είναι λοιπόν η σλιβερή κατάσταση, κατοντάδες ε, θύματα. Και στη συζήτηση ε, οπωσδήποτε θα επανέρχεται αυτό το θέμα συχνά. Λοιπόν, έχουμε πρώτο πυλώνα τρίτες χώρες, δεύτερο πυλώνα είναι τα άμεσα σύνορά μας Μεσόγειος και ο τρίτος πυλώνας είναι αλληλεγγύη και ευθύνη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαία δηλαδή της αλληλεγγύης και της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και έχω δει ε, ορισμένες, ορισμένες ομάδες έχουν περιχαρακωθεί η μεν πίσω από τη σημαία της αλληλεγγύης και η δε πίσω από τη σημαία της ε, ε, ευθύνης και δεν εκφράζονται, δεν προτείνουν τίποτα. Ε, αυτή λοιπόν η περιχαράκωση δεν ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θέλουμε να εμπεδώσουμε ναι, μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να ε, λειτουργήσει σωστά το σύστημα ασύλου, θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε επίγουσες και έκτακτες καταστάσεις χωρίς να εξωστρακίζουμε τρίτες χώρες. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σωστά να εφαρμόσουμε το άρθρο 33 και λοιπά και λοιπά. Σωστή και υπεύθυνη εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων. Ε, πρέπει λοιπόν Τώρα, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, συγκεκριμένα τώρα για την Κεντρική Μεσόγειο και τις ε, χώρες, ε, τη Λιβύη παραδείγματος χάρη και εν συνεχεία πρέπει όλοι να θέσουμε το ερώτημα τι μπορεί να κάνει ο καθένας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της ομάδας δράσης Μεσογείου αλλά και στην επόμενη πενταετία Εάν δηλαδή θα ε, βελτιώσουμε την εφαρμογή νομίμων οδών μετανάστευσης, εάν ε, μπορέσουμε να πείσουμε ε, το, τους πολίτες μας ότι εφαρμόζουμε μια σωστή πολιτική στα εξωτερικά σύνορα και ήδη φοβούμε ότι τους επόμενους δύο μήνες θα αναγκαστούμε να συζητήσουμε ε, την φρούρηση των συνόρων της Ευρώπης και το κόστος στον προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Τώρα, πώς μπορούμε το σύστημα, το όλο θέμα αυτό του ασύλου, το οποίο εσείς αποφασίσατε, να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά. Και προφανώς ε, πρέπει να συζητήσουμε εξαιρετικά δύσκολα θέματα όσον αφορά την ε, λαθρέα και παράνομη διακίνηση ατόμων. Βλέπετε λοιπόν ότι οι δράσεις στην κεντρική Μεσόγειο, οι ανταπόκριση με βραχυπρόθεσμες δράσεις, τις οποίες θα αποχρεωθούμε να λάβουμε, δημιουργούν όλο και περισσότερα ερωτήματα. Όμως, την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν τις απαντήσεις μας. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά, Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκτιμά ιδιαίτερα ε, ένα γραφειοκράτη όταν μακρηγορεί. Ε, ε, θέλω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των μελών σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Διευθυντά και ευχαριστούμε πολύ που δεν μακρηγορήσατε αλλά επισημάνατε μόνο κάποια από τα βασικά στοιχεία της ε, ειδική ομάδας για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα να ζητήσω να κάνει το ίδιο και η Ιταλική Προεδρία. Μην ε, υπησέλθετε σε λεπτομέρειες, προσπαθήστε να πείτε τι έχει γίνει, δηλαδή να εντοπίσετε τα βασικά στοιχεία ε, του, παλέ, του πακέτου του ασύλου, δηλαδή ΕΑΣΟ κλπ. Ε, τι θεωρείτε ότι, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε αυτό. Γιατί φυσικά το Συμβούλιο ε, έχει το, την αρμοδιότητα της εφαρμογής. Μη μας ε, δώσετε μας βγάλετε ένα λόγο, αλλά ε, μιλήστε επί της ουσίας γιατί πολλά από τα μέλη έχουν την εμπειρία. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Κολόμπο και ο κύριος Κάπου εκ μέρους της Ιταλικής Προεδρίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Φιλίππο Κολόμπο, συντονιστής των θεμάτων ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας στις Βρυξέλλες. Δύο λόγια θα πω μόνο επειδή η εισαγωγή που έκανε ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Ρότερ, ε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δύο λόγια μόνο για αυτά τα οποία πρόσφατα ακούστηκαν, υπόθηκαν στο άτυπο Συμβούλιο Τζάι, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Ένα πολιτικό θέμα το επόμενο διάστημα, όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής, θέλουμε να ξεπεράσουμε το θέμα του ποιος είναι υπεύθυνο για τι. Γιατί από πολλές πλευρές η συζήτηση είναι τεχνητή. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Όπως είπε για κάποιος στην Συνανδρία του Μιλάνου, υπάρχει γενική έλλειψη ικανοποίησης για το πώς έχουν τώρα τα πράγματα, για τον τρόπο με τον οποίο ε, οι χώρες υποδοχής, οι χώρες ε, μετάβασης ε, κινούνται. Υπάρχει γενική έλλειψη ικανοποίηση. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε στου επόμενου μήνε είναι να φροντίσουμε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίηση. Λαμβανωμένη υπόψη βεβαίω του μεγέθου του προβλήματο, δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα, αλλά θα σαφώ ελπίζουμε σε κάποια μέτωπα να προχωρήσουμε. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε στο να ξεπεράσουμε την αντιμετώπιση των πραγμάτων ε, ως ε, κατεπηγόντων γιατί όπως είπαν και οι υπουργοί σήμερα το πρωί η, ε, υπόθεση, η επιχείρηση Μαρενόστρουμ ε, ε, ξεκίνησε ως αντιμετώπιση μιας επίγουσας ανάγκης όταν θεωρήσαμε ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Και αυτό οδήγησε στο Μαρενόστρουμ. Πρόκειται για μια προσωρινή επιχείρηση προφανώς και ως εκ τούτου θα δώσει τη θέση της σε μια πιο βιώσιμη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών των ροών της μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η Κεντρική Μεσόγειος είναι ο χώρος με τον, την πιο εμφανή μεταναστευτική πίεση. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι όλα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα εξωτερικά σύνορα είναι ή θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν ε, αντικείμενο μεγάλων πιέσεων. Οπότε στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο όχι ε, να τυποποιήσουμε ε, την αντιμετώπιση, αλλά να καταλήξουμε σε μια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση των θεμάτων της μετανάστευσης η προσέγγιση μέσω πολλών πυλώνων που περιέγραψε ο Γενικός Διευθυντής προηγουμένως μας βρίσκει σύμφωνος και ελπίζουμε ότι πλέον θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή γίνονται τεχνικές συζητήσεις και συζήτηση μεταξύ των μονίμων προσώπων ώστε σύντομα να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης και να έχουμε και πολιτική υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Οπότε Βράχει πρόθεσμα σημαίνει αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε δράση και σε τρίτες χώρες αλλά και να επιχειρήσουμε να έχουμε δυνατότητες δράσης που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε με βιώσιμο τρόπο την τρέχουσα κρίση στην Κεντρική Μεσόγειο. Βεβαίως, όπως υπεγράμμισαν και οι Υπουργοί σήμερα το πρωί, ένα από τα βασικά ζητήματα θα είναι η ενίσχυση της Frontex. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, αν μας ενδιαφέρει να έχουμε επιχειρήσεις στην Κεντρική Μεσόγειο για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κατάσταση. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο που θα παίξει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να εμπλακεί όχι μόνο σε θέματα προπολογισμού όταν τεθούν, αλλά και πολιτικά. Να υπάρχει λοιπόν πλήρη συνέστηση σε ολόκληρη την Ευρώπη τι ακριβώς χρειαζόμαστε και τι θα χρειαστούμε στο πλαίσιο της κοινή δράσης. Όχι μόνο στο θέμα της επιτήρησης, αλλά για να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί σωστά και το Δουβλίνο. Υπάρχουν διάφορα ε, εργαλεία διαθέσιμα στα πλαίσια του Δουβλίνου και εμείς ως χώρα υποδοχής έχουμε υποχρεώσεις την ταυτοποίηση και την υποδοχή πρέπει να εγγυηθούμε οι υποχρεώσεις αυτές να τηρούνται απόλυτα. Και ελπίζουμε ότι όλοι θα θεωρήσουν ότι το Δουβλίνο τους προσφέρει διάφορες εναλλακτικέ ώστε να γίνει μια βιώσιμη διαχείριση αυτής της έντονης ροής ετούν τον άσυλο. Και όσο είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε ότι οι φιλοδοξίες των προσφύγων αυτών να ε, υλοποιηθούν, διότι μην ξεχνάμε αυτό που λέμε σήμερα το πρωί, ε, φεύγουν από καταστάσεις ε, τραγικές. Τέλος. Είναι υπάρχει ένας χώρος που πρέπει να μελετήσουμε. Είναι το τι συμβαίνει με αυτούς που τώρα βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και που φθάνουν στη Βόρεια Αφρική. Ελπίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα θα είναι δυνατόν να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας το οποίο θα ενισχυθεί και που θα περιλαμβάνει και ένα στοιχείο επανεγκατάστασης. Ελπίζουμε ότι όλοι μας θα μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο μας συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μου τέλος και πραγματικό, πραγματικά τέλος είναι το θέμα της αντιμετώπισης των ε, εγκληματιών αυτών οι οποίοι εμπλέκονται στον χώρο. Για μία ακόμα φορά. Συλλαμβάνουμε σήμερα διακινητές και ελπίζουμε ότι και σε αυτό το τομέα βραχυπρόθεσμα θα μπορέσουμε να δράσουμε πιο εντατικά ότι θα έχουμε τα μέσα να το κάνουμε και ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών και με τη χρήση των επιτόπου δικτύων, ώστε να κινηθούμε ταχύτατα και να συλλάβουμε τους διακινητές της σε τρίτες χώρες της δικές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω στα νέα μέλη ε, που ε, έχουν πρωτοέρθει ότι η Προεδρία έχει την ευθύνη του να καθοδηγήσει το πρόγραμμα δράσης, ενώ το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να κάνει αυτό που έχουν κάνει εδώ πολλά μέλη, δηλαδή το πακέτο του Δουβλίνου, τα, στο, για το οποίο έχουν συμμετάσχει με τη δουλειά τους και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να διαγνώσουμε πως έχει η κατάσταση ε, στους διάφορους τομείς. Το πρόβλημα είναι η υλοποίηση. Αυτό συζητήθηκε στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ισοτορικών. Κάποια νομοθεσία δεν υλοποιείται και αν οι οργανισμοί δεν έχουν αποτελεσματικό έργο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να διαγνώσει την κατάσταση. Ενημερώνω για όλα αυτά τα νέα μέλη. Έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο διάφορα μέλη. Παρακαλώ να λέτε το όνομά σας. Σίπολ, Κάρακολ. And then members, Mr. Diaz de Mera, uh, Mrs. Gomez, Mrs. Daly, um, uh, Ska Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Υπάρχει άλλος που θα ήθελε το λόγο? Κύριος Κύρκος. Έχουμε πολύ χρόνο. Yeah, and we've got, um, if you stick to... Yeah. Ε, είπα κάτι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη που είπα ότι έχουμε πολύ χρόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ύστερα από τον εφιάλτη που ζήσαμε σήμερα το πρωί, πιστεύω ότι τώρα θα τα καταφέρουμε υπάρχει και ισότητα, οι συντονιστές θα πάρουν τον ίδιο χρόνο. Θα έχουν τον ίδιο χρόνο όπως και όλοι οι άλλοι. Θα υπάρξει ισότητα και έχετε χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Δύο, λεπτά περίπου. Περίπου δύο λεπτά ο καθένας σας, παρακαλώ. Να... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο λεπτά περίπου ο καθένα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα δύο λεπτά. Είπατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις 300 διαφορετικές δράσεις. Άρα το θέμα μετανάστευση, η κατάσταση στη Μεσόγειο προσεγγίζεται με πολλές διαφορετικές ε, απόψεις και με πολλές διαφορετικές οδούς. Όμως πολλές φορές και επανειλημμένα ακούγεται η άποψη ότι η Frontex θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Η Frontex όμως είναι η υπηρεσία προστασίας των συνόρων. Δεν έχει σχέση με το μεταναστευτικό. Τι εννοούν λοιπόν όταν λένε πρέπει να ενδυναμωθεί, να, πιο, να γίνει πιο πυκνή η φρούρηση των συνόρων. Όμως τι θα γίνει τότε με τους πρόσφυγες που θέλουν να μπουν μέσα. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που δικαιούνται να ε, μπουν στο, στην επικράτειά μας, ότι είναι γνήσιοι πρόσφυγες και διώκονται για πολιτικούς λόγους, ε, ε, ότι θα μπορέσουν να μπουν και να ζητήσουν άσυλο. Το δεύτερο θέμα, πολλοί πρόσφυγες δεν είναι πρόσφυγες λόγω συγκρούσεων ε, και πολέμων αλλά λόγω οικονομικών δεινών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ε, τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις θέσεων εργασίας σε ορισμένους ε, τομείς για να δοθούν ορισμένες ευκαιρίες νόμιμης μετανάστευσης για οικονομικούς μετανάστες. Και τρίτον το θέμα του πακέτου μέτρων για το άσυλο. Για το άσυλο. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση μέτρων που προβλέπει αυτό το πακέτο που έχουμε, το οποίο έχουμε αποφασίσει. Και τελευταίο ζήτημα το Δουβλίνο, η κατανομή των προσφύγων και η εθελοντική υποδοχή ποσοτική υποδοχή δηλαδή προσφύγων. Μπορούμε να πούμε, να υποθέσουμε ότι αυτά όλα θα εφαρμοστούν σωστά στο προσεχές με άλλο που θα αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων. Ευχαριστώ Μπριγκίτε. Μπορείτε να εκφράσετε βέβαια κάτι που ξέχασα να το πω, όχι μόνο τι ερωτήσει, αλλά και κάποια γενική τοποθέτηση. Πολλοί από εσά άλλωστε είναι ιδιαίτερα έμπειροι. Μπορείτε να δώσετε λοιπόν την άποψή σα Δεν ε, είναι απαραίτητο να περιουστείτε σε ερωτήσεις. Θα προσθέσω και τη συνάδελφο που κατά λάθο δεν σας έδωσα το λόγο το πρωί και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κέρκοπ για την ομάδα ECR που είναι ο συντονιστής. Κύριε Πρόεδρε, καταρχά θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά και ισχύει για όλους φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας γιατί και εγώ προσωπικά έχω δεχθεί πέσει, αλλά και όλοι δεχόμαστε καθημερινά ε, πιέσει και έχουμε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση λόγω των ε, ισρώων. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε Είναι σαν να βάζουμε απλά ένα επίδεσμο ε, σε μια μεγάλη πληγή, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την αναλογία. Πάρα πολλά άτομα έφτασαν στα κτές της Ιταλίας και αναμένονται ακόμη περισσότερα. Με την ισχύ που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται, να, ε, θα έπρεπε να ισχύει μια πιο κοινή προσέγγιση, πιο συντονισμένη προσέγγιση. Σίγουρα η Ιταλία υποδέχεται μεγάλο αριθμό ατόμων, όμως Επίσης, σημαντικό μέρος αυτών δεν παραμένουν στην Ιταλία. Οι όροι και οι συνθήκες τις οποίες φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και όσοι πλέον ε, ευνοϊκές ε, Ίσως ο σεβασμός δεν είναι ο κατάλληλος, διαδικασίες ε, που εφαρμόζονται για την καταχώρησή τους, ε, για να ενημερώνονται κτλ. Ίσως να μην είναι και οι πλέον κατάλληλες. Θα έπρεπε λοιπόν ε, να δούμε περισσότερο τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας στις χώρες προέλευσης, καταγωγής ή ίσως, ίσως τις όμορες αυτών χώρες, να φροντίσουμε οι συνθήκες να είναι καλύτερες, να δοθούν περισσότεροι πόροι όπου δει και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Θα μπορούσαμε και με τα Ηνωμένα Έθνη να συνεργαστούμε. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε αντί απλά να αντιμετωπίζουμε, να διαχειριζόμαστε καταστάσεις ε, που σίγουρα θα επιδεινωθούν, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά ε, των διακινητών, και να δούμε ποια είναι τα κίνητρα και για ποιους λόγους εγκαταλείπουν τις χώρες τους υπό αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα δεν έχει άμεση ευθύνη για τους πρόσφυγες η Frontex, ωστόσο η Frontex όλο και περισσότερο αντιμετωπίζει στη θάλασσα αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχουμε λάβει ε, παρκώ σοβαρά το θέμα, ούτε έχουμε διαθέσει επαρκή πόρου και μέσα. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί κύριε Πρόεδρε, η δύσκολη προς το παρόν πρόκληση μπορεί να γίνει ένα πραγματικό χάος στο μέλλον, να έτσι φοβούμε και αυτό θα ήταν κακό για τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ολόκληρη την Ευρώπη βέβαια. Πρόεδρος, η Σεσίλια Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, που φυσικά και έχει ζωτική σημασία και πρέπει να συνεχίσει η ειδική ομάδα και το έργο της πρέπει βέβαια να φέρει απτά αποτελέσματα. Και επειδή φαίνεται ότι για να φτάσει κανείς στο ευρωπαϊκό έδαφος ε, αντιμετωπίζει κανείς σχεδόν ε, πάντα ε, δυσκολίες, νομικές και άλλες, ε, πολλές φορές πέφτουν θύμα αυτοί οι άνθρωποι διακινητών και γίνονται παράνομοι μετανάστες μέχρι να φτάσουν καταθέσουν αίτηση ή τη χορήγηση του καθεστώτος ασύλου σε μια χώρα. Με ανησυχεί λοιπόν, με ανησυχεί η γλώσσα, οι διατυπώσεις που βλέπω στη σελίδα 3 για παράδειγμα για το δίκτυο που λέει ότι το δίκτυο καταπολεμά Shall Combat ως υποχρέωση την λαθρομετανάστευση. Αλλά πώς καταπολεμούμε τη λαθρομετανάστευση όταν δεν φροντίζουμε να υπάρχουν ασφαλείς διάδρομοι και νομικές ευκολίες προς αυτά τα άτομα. Φυσικά και θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάστευση αλλά και να σώσουμε ζωές ταυτόχρονα. Άρα πώς θα πετυχαίνουμε αυτά τα δύο εάν έχουμε ε, ε, ασφαλείς και νόμιμες οδούς ε, προς την ε, Ένωση. Σε μια παράγραφο λέγεται ότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, την νόμιμη πρόσβαση στην Ένωση. Και έπειτα ε, γίνεται λόγος αυτή την παράγραφο για τη μετανάστευση και διάφορα άλλα θετικά. Εγώ είμαι εισηγητρία για τους φοιτητέ και τους ερευνητές, για τους οποίους επίσης γίνεται λόγο στην παράγραφο αυτή και καλό θα ήταν σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία υπήρξα και και για, την, ε, για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ξέρω πολύ καλά περί πρόκειται λοιπόν. Για αυτούς όλους τους λόγους πιστεύω θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρέπει να βρούμε να δώσουμε δυνατότητες ε, ώστε οι ετούντες άσυλο νομίμως να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς ε, οι διακινητές θα συνεχίσουν να μεταλλεύονται αυτά τα άτομα και να είναι συνεχώς σε κίνδυνο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλός, γελία χαμηλός θα έλεγα ο αριθμός των χωρών ε, που συμμετέχουν και των ανθρώπων που υποδέχονται. Κάποια κράτη δεν συμμετέχουν δε καθόλου. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση για την επαναγκατάσταση. Μαζί με την Υπατιαρμοστή για τους πρόσφυγες και την ε, Επιτροπή μπορείτε να προχωρήσετε με το θέμα αυτό της επαναγκατάστασης και το θέτω και στο Συμβούλιο το θέμα, γιατί είναι στα χέρια του Συμβουλίου, που πρέπει πλέον να υπογραμμίσει τη σημασία των τεκτενωμένων στη Μεσόγειο και στα κράτη-μέλη, συγκεκριμένα στο δικό σας, στην Ιταλία δηλαδή, ώστε τελικά και επιτέλους να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το αίτημά μας. Δεν θέλω να σας τριμώξω στη γωνία, σε καμία περίπτωση, απλά θέλω να σας δείξω ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό και να μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε και να βρούμε τρόπους να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να λάβουν τις ευθύνες τους και να δείξουν υπευθυνότητα. Επίσης, επικροτώ και την έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων σε πρεσβείες των ομεθνών ή σε προσωρινά ε, προξενικά γραφεία στους καταβλισμούς. Αυτό σίγουρα θα σώσει ζωές και λυπούμε και θέλω να το τονίσω ότι δεν αναφέρεται καθόλου αυτό το μέτρο στο έγγραφο για την ειδική ομάδα. Γιατί αυτό το τόσο σημαντικό θέμα αποσιωπάται εντελώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, Σεσίλια. Κύριο Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να καλωσορίσω τον κύριο Ρούτε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία με τον προκάτοχό σας είχαμε μια καλή επικοινωνία και σήμερα το πρωί μόλις του έγραψα, ε, μάλλον σας έγραψα μια επιστολή και σας ζήτησα συνάντηση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά αλλά και την Επιτροπή μας. Έξω και δεν θα σας κάνω κάποια ερώτηση κύριε Ρούτε, θα ακολουθήσω τις ε, συστάσεις του Προέδρου Κλοντ Μωράης, επομένως θα περιουστώ σε κάποιες σκέψεις γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου για να σας εξηγήσω εδώ και τώρα αναλυτικά τις απόψεις μου. Όπως λέει και ο τίτλος του σημείου αυτού της ημερήσιας διάταξης, ο λόγος είναι ακριβώς η ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο. Δεν καλύπτει άλλα θέματα το σημείο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σύμφωνο σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η Σεσίλια Βίκστρομ μόλις τώρα. Πραγματικά ε, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα αυτά που είπε, διότι Υπάρχει και ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ότι σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και επειδή είναι επίκαιρα, πολύ επίκαιρα όλα αυτά, στη Μεσόγειο, κύριε Ρίτε, έχουμε την Ανατολική Μεσόγειο που εκεί είναι οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις. Υπάρχει όμως και η Κεντρική Μεσόγειο έχουμε αυτή την τραγωδία εκεί, λιγότερες μεταναστευτικές πιέσεις από ό,τι στην Ανατολική και έχουμε και τη Δυτική Μεσόγειο που έχουμε επίσης τραγωδία στα χερσαία σύνορα στη Βόρεια Αφρική και στις ακτές της Ισπανίας. Η Frontex ανέλαβε κάποιες δράσεις για τον ελέγχο συνόρων. Έγιναν λοιπόν, ανέλαβε μια σειρά από επιχειρήσεις. Χρήσιμες και απαραίτητες θα έλεγα. Δεν αρκούν όμως. Είναι σαφές όμως ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι πρέπει να ενισχυθεί η Frontex. Και γιατί διότι η εμπειρία μου μου έχει διδάξει ότι τεχνικός πως είναι αδύνατο να μπορεί κανείς ε, χιλιάδες χιλιόμετρα ε, θαλάσσης να μπορεί κανείς να τα επιτηρεί συνεχώς για να προστατεύει τα σύνορα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. επιχείρηση Mare που είναι άλλωστε και η διαπίστωση της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η απάντηση στην ε, αποτυχία ε, που χαρακτήρισε την επίγουσα δράση της Ένωσης. Αν κάτι έχει να μας διδάξει ή χρησιμεύει κάτι αυτή η επιχείρηση Μάρι Νόστρομ, δεν είναι η προστασία των συνόρων, ξέρετε. Είναι η διάσωση ανθρώπων. Το να σώσει ζωές, αυτό το στόχο έχει αυτή η επιχείρηση. Καλή και ε, επιτυχημένη από αυτή την έννοια και καλή και ενίσχυση της Frontex αν είναι αυτός ο στόχος. Γνωρίζουμε όμως ότι η Frontex είναι συνεργασία και ξέρουμε ότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Τι κάνει η Frontex λοιπόν. Η Frontex είναι η διαπίστωση του ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι και κοινά και πρέπει να τα προστατεύσουμε, να τα περιφρουρήσουμε. Για ποιο λόγο. Για να προστατεύσουμε μία από τις σημαντικές ελευθερίες που εμείς ορίσαμε και που είναι η ελευθερία διακίνησης, διέλευσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Πρόσφυγες, άσυλο, όχι. Δεν έχει ακόμη η Ευρώπη κοινή πολιτική σε θέματα ασύλου. Δεν είναι αλληλέγγυα η Ευρώπη σε θέματα ασύλου. Ούτε ισομερός και δικαίως ε, ε, επιμερίζει ε, αυτό που λέμε επιμερισμό βάρο επιμερίζει τον αριθμό των ε, ε ετούντων άσυλου. Η Βουλγαρία, το ακούσαμε. Μπορεί η Βουλγαρία μόνη της να δεχθεί όλους τους πρόσφυγες από τη Συρία ή από τη Λιβύη. Όχι. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια πραγματική και αλληλέγγυα πολιτική ασύλου. Αυτές είναι λίγες από τις πολλές μου σκέψεις για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η ευρωπη πρεπει επιτελους να αποκτησει μια πραγματικη και αλληλεγγυα πολιτικη ασυλου αυτες ειναι λιγες απο τι πολλε μου σκεψει για αυτα τα θεματα ευχαριστω ο ευχαριστω η βουλγαρια και η Σουηδία ήταν τα δύο παραδείγματα για το, στο Συμβούλιο Τζάι για τη Συρία όταν μιλήσανε. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Σκάλ Κέλλερ. Ε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στο καινούριο σας πόστο, η καινούργια σας δουλειά κύριε Ρίτκε. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τέθηκαν, τα έχουμε πει ξανά και ξανά και ξανά και ε, ερωτήματα προς την ομάδα δράσης ε, για την Μεσόγειο είναι αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε. Οι δράσεις αυτές που αναφέρετε είναι αυτές που προτείνονται, είναι ορισμένες που ήδη εκτελούνται ή πρέπει να εγκριθούν για το μέλλον τι γίνεται με αυτές τις 200 και δράσεις. Και από την πλευρά των πρασίνων ένα από τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε και το έχω πει και οι φιλελεύθεροι, όπως είπαμε και το, όπως μάλλον δεν ελέγξει το πρωί ε, με την Ιταλική Προεδρία διότι ο, Ιτα, ο Ιταλός, ε, η Ιταλική Προεδρία δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας ε, που θέσαμε για τους πρόσφυγες και τους, ε, το μεταναστευτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι οδοί ε, νόμιμης ή παράνομης μετανάστευσης. Εμείς θέλουμε να έχουμε νόμιμη μετανάστευση. Πολύ ωραία και σωστά η η για τους πρόσφυγες λέει ότι η μετανάστευση λοιπόν πρέπει να είναι μία και ε, η ύπατη αρμοστή βεβαίως κοιτάει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των νομίμων προσφύγων. Έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες, ε, ε, σκοπιμότητες, αναλύσεις και όλα αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά. Πώς μπορούμε τώρα λοιπόν από, αφενός να λύσουμε το πρόβλημα του, του, του δράματος που συμβαίνει και αφετέρου να εξασφαλίσουμε ότι παραμένουν ανοιχτές οι, οδοί, οι δρόμοι, ανοιχτοί οι δρόμοι της νόμιμης μετανάστευσης. Το έχει πει και ο Πρόεδρος και άλλα μέλη. Τι θέλετε η Frontex να κάνει. Πολλοί λένε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Frontex κλπ. αυτό η Frontex αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά προβλήματα από ότι πρόσφυγες ας πούμε τη Συρίας τι ακριβώς θέλετε για τη Frontex. Επιπλέον εκατομμύρια, εκτός από τα πολλά εκατομμύρια τα οποία ήδη λαμβάνουν, τη χρηματοδότησή τους δηλαδή, τι θέλετε ακριβώς για τη Frontex. Θα, επιτέλους, θα, θα, θέλαμε να ξέρουμε την άποψή σας, διότι μπορεί και να συμφωνήσουμε. Κάθε φορά λέγεται το, το είναι ενισχύστε τη Frontex, αλλά δεν ξέρουμε τι, τι εννοείται και τι χρειάζεται. Επίσης το Δουβλίνο, ακούγεται ότι το Δουβλίνο, η συμφωνία του Δουβλίνου πρέπει να βελτιωθεί κλπ. κλπ. Πώς ακριβώς, ε, τι εννοείται με τη βήματα, τις συγκεκριμένε ενέργειες. Ποια είναι η κατάσταση τώρα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Θα προτείνει η Κομισιόν νέες πρωτοβουλίες για το Δουβλίνο. Ο πρόεδρος, η, κυρία Νταλή, η Μίριαμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερόμενους ε, που έχουν εκφράσει απόψεις για την υλοποίηση των μέτρων και την, την ομάδα εξωτερικής ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι συναρμόδιοι θα πρέπει ε, επιτέλους να υλοποιήσουν τα μέτρα της ομάδος δράσης. Και αναφέρουμε στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης του, και του οργανωμένου εγκλήματος. Και επίσης να ταυτοποιήσουν επιτέλους αυτά όλα τα ε, δίκτυα, τα παράνομα δίκτυα είτε αφορά, ε, αναφέρουμε στην Κομισιόν, στην EAS, Ομάδα Εξωτερικής Δράσης, στην Frontex, εάν δεν υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα δεν ε, προσθέτουν, ε, δεν προσφέρουν πρόσθετη αξία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλή εφαρμογή όλων αυτών των ε, προσπαθειών με, με πρωτοβουλίες, με επιπλέον πρωτοβουλίες. Και ε, πρέπει να δράσουμε διότι μέτρα τα οποία προβλέπονται υπάρχουν ήδη και πρέπει να δράσουμε επιγόντως διότι έχει δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Ε, και θα θέλω αυτά τα πολιτικά προγράμματα επιτέλους να αρχίσουν να εφαρμόζονται διότι ο χρόνος έχει πλέον οριμάσει. Και ε, πιστεύω ότι το πρόγραμμα για την ενίσχυση της γρηγορότερης εξέτασης των προσφυγών ασύλου έχει ήδη λειτουργήσει, είναι, εκτελείται ήδη και θα ήθελα η Κομισιόν να μας πει, ε, να μας ενημερώσει για το τι άλλες δράσεις θα λάβει σε αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Γκόμες. Ακόμα και αν η προσέγγιση Ακόμα και αν η προσέγγιση είναι ε, γραφειοκρατική, μου φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική είναι κάπως ε, είναι ουτοπική δεν είναι ρεαλιστική, διότι βασίζεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτό δεν θα επιτύχει. Εάν όλα μας τα όργανα της εξωτερικής πολιτικής καταλήγουν σε αποτυχία. Δηλαδή, όλες αυτές τις συμφωνίες επαναπατρισμού και επαναπρόθεσης δεν λειτουργούν. Για, για ποιο λόγο να συζητούμε τη Λιβύη και οι ηγέτες μας μιλάνε και αναφέρονται συνέχεια για τη Λιβύη λέγοντας ότι είναι μια χώρα σταθής. Αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα πλήρως αποτυχημένη και ε, στο προηγούμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ζήτησαν οι Υπουργοί παρέμβαση για να ε, αποφύγει η Λιβύα με πλήρη κατάρρευση και τα άτομα τα οποία έρχονται μέσω Λιβύης είναι άτομα από όλες τις χώρες της Αφρικής. Κοιτάξτε τι γίνεται στο κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, στην Αιθιοπία, στο κέρας της Αφρικής. Από εκεί προέρχονται όλοι αυτοί που προσπαθούν να περάσουν απέναντι μέσω Λιβύης. Λοιπόν, τι νόημα έχει να μιλάμε με γενικότητες και με ουτοπικά, ουτοπικές ιδέες. Πρέπει επιτέλους να συνέλθουμε και να γίνουμε ρεαλιστές και να εφαρμοστεί επιτέλους η εξωτερική μας πολιτική. Διαφορετικά ε, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και τίποτα δεν θα επιτύχει. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η επίπτωση αυτών των μέτρων λιτότητος στους εθνικούς μας πόρους και στην δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις και να κάνουν αυτά τα οποία είναι αναγκαία. Εγώ σκέφτομαι τη δική μου χώρα, την Πορτογαλία. Παρόλο που υπάρχει βούληση των αρμοδίων, δεν έχουν τους πόρους. Υπάρχει μια μεγάλη κρίση διαθέσιμων πόρων και όλες οι υπηρεσίες ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα βρίσκονται σε δινή θέση. Εάν λοιπόν ε, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και αν θέλουμε να επικεντρώνουμε και να, ενισχύσουμε την νόμιμη μετανάστευση πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλύτερη δουλειά από αυτή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η Σιλβή. Dans ε, θα επαναλάβω με διαφορετικό τρόπο αυτό που είπε η Άννα. Αυτή η ειδική ομάδα δράσης Μεσόγειος ε, είναι κάτι το οποίο συνεχίστηκε μετά από την πρώτη τραγωδία της ε, Μεσογείου και η ίδια η Επίτροπος Μάλμστρομ το παραδέχθηκε σε κάποιο έγγραφο ότι δεν, προσφέρει, δεν προσφέρει κάτι το καινούριο. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι για μία ακόμα φορά πρέπει να ξέρουμε, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση αυτών, των, αυτών, αυτών, αυτών τα οποία γίνονται. υπάρχει ένας ε, κατάλογος ε, πραγμάτων που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη και να μην πρέπει να εφαρμόζονται αυτά με τρόπο στερητικό της ελευθερίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παρακινηθούν τα κράτη-μέλη να ε, λάβουν μέτρα που είναι λιγότερο δημοφιλή όπως η επανεγκατάσταση ας που αναφέρθηκε, η ανθρωπιστική βίζα ή η προστατευόμενη είσοδος. Πρέπει, κανείς να, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά. Το τρίτο θέμα που θέλω να φερθέρω και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά γνωρίζετε ένα σχέδιο που ονομάζεται MOAS, Migrant Offshore Aid Station, που από ό,τι άκουσα υποτίθεται ότι θα, είναι, θα αποτελεί επιχείρηση ε, διάσωσης ε, που χρηματοδοτείται από ιδιωτικού πόρους. Πρόκειται ε, για μια πρωτοβουλία ενός ζευγούς από τη Μάλτα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αστείο ή φάρσα ή κάτι άλλο. I heard about Έχω ακούσει κάτι αλλά δεν ξέρω. Η Μαρία μπορεί να... Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν σας δίνω τώρα το λόγο. Κάτι έχω ακούσει, κάτι κυκλοφορεί από αυτό αλλά ίσως οι συνάδελφοι από τη Μάλτα να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα από αυτού. Επόμενος ομιλητής, μακραίνει ο κατάργος των ομιλητών και φταίω εγώ που είπα ότι υπάρχει πολλής χρόνος. Ο κύριος Κύρκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δύο προηγούμενοι συναδέλφοι έθεσαν το θέμα πάρα πολύ στην καρδιά του και δεν έχω να προσθέσω πολλά. Απλώς ότι όπως βλέπω για την Ιταλία, αλλά σίγουρα για την Ελλάδα, η Frontex και η Task Force προσφέρει ε, και συμβάλλει ουσιαστικά στο να αποφευθούν τραγωδίες στη θάλασσα. Ε, όμως, για να ε, συμβεί αυτό καλύτερα, οι δράσεις της Task Force θα πρέπει να επεκταθούν ουσιαστικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην επικεντρώνονται μόνο στην Κεντρική Μεσόγειο ή κυρίως στην Κεντρική Μεσόγειο. Βεβαίω αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πίεση μετανάστευση προέρχεται από την υποσαχάρη Αφρική και από τη Λιβύη. Όμω οι μεταναστευτικέ ροέ εξελίσσονται δυναμικά. Ε, με τη Συρία, με το Ιράκ, με την Παλαιστίνη βλέπουμε ότι αυξάνεται σημαντικά ο ρυθμός των ε, προσφύγων οι οποίοι έρχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε θα είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το σύνολο της Μεσογείου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα την άποψή σα, εάν συμφωνείτε, και αν είναι με συγκεκριμένες δράσεις θα εκφραστεί αυτό. Επίση, η, η μεγαλύτερη δέσμευση τρίτων χωρών σε ενημερωτικέ εκστρατείε και στα προγράμματα περιφερειακή προστασία είναι απαραίτητη ώστε οι μετανάστες να είναι ενήμεροι για την ε, παράνομη δραστηριότητα των διακινητών και τα επικίνδυνα για τη ζωή του ταξίδια. Μέχρι στιγμή, τα προγράμματα αυτά δεν απευθύνονται στι χώρε τη Ασία, από όπου και υπάρχει ισχυρή μεταναστευτική ροή. Ε, υπάρχει σχέδιο να συμπεριληφθεί και η Ασία τελικά σε αυτά. Ευχαριστώ. Uh, ο Τόμας Τετόφσκι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτερ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Είμαι ειδικό σε θέματα στρατηγικής και ως εκ τούτου θα ήθελα να μάθω υπάρχει κάποια στρατηγική και ποια είναι ακριβώς τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ιταλία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας τίποτα. Διότι αυτό το οποίο μου φαίνεται ότι λείπει είναι η στρατηγική. Ευχαριστώ. Μας εκπλήξατε. Μας εκπλήξατε μιλώντας ιταλικά ορισμένοι μείναμε λίγο. Τέλος πάντων, επόμενος ομιλητής. Βίμπερ. Διαλέξτε εσείς τη γλώσσα θα χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μεσόγειο είναι πραγματική τραγωδία, άνθρωποι οι οποίοι πνίγονται προσπαθώντας ε, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και αυτό είναι πολύ καλό. Το ερώτημα είναι όμως πώς. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι με την αύξηση των πόρων και μέσων της Frontex ε, θα σώσουμε ζωές, θα ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα ίσως χάσουν και το ενδιαφέρον τους οι διακινητές και πάψουν να ασχολούνται τόσο με την εμπορία ατόμων, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε νωρίτερα η Σεσίλια Βίκστρομ. Ο κόσμος που προσπαθεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε επιλεκτικοί ποιον θα αφήσουμε να μπει και ποιον όχι. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω τις σκέψεις σας. Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει επιτόπου να παράσχουμε βοήθεια και στους καταβλισμούς προσφύγων, κυρίως μέσω της ΥΠΑ Αρμοστίας. Βέβαια έχουμε και τη σύμβαση του Δουβλίνου. Εγώ είμαι Σουηδέζα και βλέπω στη χώρα μου να υπάρχει αναβλητικότητα από κάποιες μεσογειακές χώρες. Βέβαια υπάρχουν ψηλέ πιέσεις. Στη Βόρεια Ευρώπη βιώνει αυτές τις πιέσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές και σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να ενταχθούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Πολλές απόψεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά σίγουρα πρέπει επιτόπου κατ' πρώτα να εστιάσουμε. Ε, τελευταίοι Βόιτ, ορίστε. Και Σάρα θα μιλήσετε κι εσείς, γιατί δεν πήρε το λόγο τελευταία φορά. Και Σεσίλ και Άγγι. Okay? Κλείνει ο κατάλογος. Επομένως. Χάλο Άχο, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου στο όνομα της αλληλεγγύης και για την αποθάρρυνση της επιλογής ε, ε, χώρας ε, για την κατάθεση της ασύλου, asylum shopping όπως το έχουμε αποκαλέσει. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικούς κανόνες σε ό,τι αφορά την ε, παροχή ασύλου ή τα οικογενειακά επιδόματα κτλ. Άρα με τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ε, ορισμένα κράτη θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τα δικά τους πρώτους δικούς τους κανόνες ή άλλα κράτη να χαμηλώσουν ε, αυτά τα πρότυπα, αυτά τα στάνταρτ. Κάτι το οποίο από πολιτική αλλά και οικονομική πλευρά, για να μην πω ότι είναι αδύνατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον. Κάτι ακόμη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλοί ε, από αυτού που έρχονται από τη μία όχθη τη Μεσογείου στην άλλη, πολλέ φορέ δεν εντάσσονται στην κατηγορία των προσφύγων, να ζητούν άσυλο, ε, γιατί δεν μπορούν να βρουν κάποιο άλλο, κάποια άλλη οδό κάποιο, για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίμως. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Η Ευρώπη, η οποία ήδη ε, πλήττεται από μια καταστροφική ανεργία, δεν έχει μέσα, δεν μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας σε χιλιάδες ανειδίκευτα άτομα ή να τα εντάξει στην κοινωνία. Την αποτυχία αυτή τη βλέπουμε, βλέπουμε και τα αποτελέσματά της σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη σήμερα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μακροπρόθεσμα, ποια είναι η στρατηγική μας. Είναι σαφές ότι η μετανάστευση ε, σίγουρα ε, δεν θα εκριζώσει τη φτώχεια από την Αφρική, ενώ από την άλλη πλευρά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τώρα θα είμαι αυστηρότερος, γιατί πέρασε η ώρα μας και πρέπει να σας σταματώ στα δύο λεπτά. Σεράια eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα ότι έγινε πιο μακρύς ο κατάλογος ε, των ομιλητών. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη λοιπόν. Τι θα επιλέξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα, είμαστε, θα δείξουμε ανθρωπισμό ή θα προσπαθούμε απλά να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Ποιος θα λάβει αυτή την απόφαση. Δεν πρέπει να τοποθετηθούμε επ' αυτού και πρώτα να γίνει αυτό και μετά να χαράξουμε στρατηγικές ή να διαθέσουμε κονδύλια στον ένα τον άλλο φορέα. Η Κριστίν Βίμπερ είπε ότι πρέπει να βοηθήσουμε επιτόπου. Δεν αποκλείω όμως το ένα το άλλο και εγώ νομίζω ότι πρέπει να δεχθούμε το γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους ε, που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν ε, τη δίωξη κτλ. Ε, Στην περίπτωση των Ρωμά, για παράδειγμα, στη Σουηδία. Αυτό που λέει το κόμμα της κυρίας Βίμπερ και η ρατσιστική του προπαγάνδα δεν ταιριάζουν ε, με την πάρα πολύ ωραία εικόνα που παρουσιάζει για τη Σουηδία και πόσο υποδέχεται πρόσφυγες κτλ. Βόητο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Και άξιο προσοχή τον κύριο Ρόιτερ. Αναφέρεται τη συμφωνία του Δουβλίνου, του Δουβλίνου και την πρώτη υποδοχή ε, είπατε ότι μπορούμε να βρούμε κάποια προσωρινά μέτρα, ότι η δύναμη κρούση, η task force έχει τη δυνατότητα να σώσει ανθρώπινη ζωή, αλλά ε, αφενός μία λύση είναι η ενίσχυση των συνόρων, η άλλη λύση είναι η νομιμοποίηση, η νόμιμη, οδο, η νόμιμη οδός. Απ' την άλλη πλευρά, ο Υπουργός σήμερα το πρωί δεν ανέφερε καθόλου μια ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή, να καταπολεμήσουμε τα αίτια της παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει να αντιπαραθέσουμε κάτι στην, στα αίτια αυτά. Δηλαδή, να μην χρειάζεται η φυγή ε, από τα εδάφη καταγωγής των ανθρώπων αυτών με λίγα λόγια δηλαδή καταπολέμηση της φτώχειας, καταπολέμηση της ε, ένδυας, ε, επενδύσεις σε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα. Αντί να μιλάμε λοιπόν συνέχεια για τη μετανάστευση, ε, μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να ξεκινήσουμε από εκεί να προσπαθούμε να κάνουμε, να καλυτερεύσουμε ε, τα δεδομένα στην πηγή ε, της δυστυχίας, δηλαδή στην, ε, στις χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύω ότι θα μέναν στις χώρες τους αν είχαν κάποια προεπτική διαβίωσης. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ η Σισίλ. Θα ήθελα να επανέλθω σε μια προηγούμενη ερώτηση που δεν απαντήθηκε ικανοποιητικά το πρωί. Όταν μίλησα για την διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου και την υποδοχή των ατόμων, αναφερόμενο, στο πώς μπορούμε να αποφύγουμε το οργανωμένο έγκλημα, την, το ξέπλυμα χρήματος και τη διαφθορά. τι προτάσεις υπάρχουν στο τραπέζι που μπορούν να εφαρμοστούν από τη δύναμη δράσης, από το Task Force. Και επιμένω σε αυτό διότι υπάρχει κάποια σύγχυση. Από τη μία πλευρά μιλάμε για την ενίσχυση της Frontex, δηλαδή ενίσχυση των ελέγχων και όχι τόσο ε, το να σώσουμε ζωές. Εάν τώρα η Frontex ενοποιηθεί με την ε, Mare Nostrum, Θέλω πιο, πολλές, ε, πιο μεγαλύτερη ενημέρωση, διότι το Μάρια Nostrum έχει πιο διευρυμένες δυνατότητες, η Frontex είναι για τα σύνορα. Η πρότασή μου λοιπόν θα ήταν ότι σε ορίσεις ε, διεθνούς ε, εφαρμογής θα πρέπει να διεθνούς ισχύως θα πρέπει να δίνονται ε, και έτσι σίγουρα θα καταπολεμηθεί μια πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει βεβαίως να αποφευθούν ε, αυτές ε, οι θεωρήσεις από το να πέσουν στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος τα οποία πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος έχουν εισχωρήσει πια παντού, παντού σε κάθε διαδικασία που ξέρουμε. Ο Πρόεδρος, Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν να μας απαντήσει σε 2-3 λεπτά για να μας πει περισσότερα για την ομάδα δράσης. Και βεβαίως ε, δεν ε, πιστεύω ότι μπορείτε να απαντήσετε σήμερα σε όλα αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε ορισμένα ζητήματα. Αλλά όπως είπε ο κ. Δίας Δεμέρο, ε, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να ξεκινήσουμε μια σχέση συνεργασίας όπως είχαμε με τον προκάτοχό σας διότι πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν και είναι σημαντικό για μας να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και δεύτερον, πρέπει να αρχίσουμε νωρίς, ε, ε, στην αρχή της ε, θητείας μας, της εντολής μας. Και γι' αυτό ακριβώς σας καλέσαμε σήμερα και είμαστε πολύ ευτυχείς που σας έχουμε σήμερα εδώ και θα σας βλέπουμε συχνά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και κάτι άλλο, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Θα επαναφέρω το θέμα αυτό στους συντονιστές μας για, τις, για τη στρατηγική. Το Σεπτέμβριο θα γίνει η συζήτηση του συντονιστές. Αυτός είναι, αυτή είναι η διαδικασία σε εμάς το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και ε, ε, με προκαταλάβατε. Ε, κατάλαβα κάτι στους πρώτους δύο μήνες της ε, εργασίας μου είναι ότι το μεταναστευτικό σε τον κύβο του Ρούμπικ το γυρίζει, το γυρίζει από εδώ και από εκεί η μία πλευρά τη φτιάχνεις, οι άλλες δεν φτιάχνονται. Μετά φτιάχνεις την άλλη πλευρά και χαλάνε οι υπόλοιπε. Λοιπόν, έτσι είναι η ιστορία. Πρέπει να Έχουμε βραχυπρόθεσμες, μέσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές και πιστεύω ότι θα, ήταν για, μένα λίγο υπεροπτικό να αρχίσω να απαντώ σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εγώ περισσότερο μίλησα μέσω και μακροπρόθεσμα, δηλαδή για την προσέγγιση αυτή. Ελπίζω την επόμενη φορά να μπορέσω να απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Ε, και ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα. Προσβλέπουμε μεγάλη ε, χαρά ε, την ε, μελλοντική μας συνεργασία. Γενικά, η μετανάστευση και η νόμιμη πτυχή της μετανάστευσης, η Σεσίλια Μάλστρομ, από πέρσι ήδη προσπαθεί να προχωρήσουν μερικά πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουν γίνει συγκεκριμένες συζητήσεις και ε, αν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μερικά από αυτά τα προγράμματα, παραδείγματο χάρη κατανομής, να βρούμε μια κλίδα κατανομής. Ίσως δεν είναι ιδανική απάντηση αυτή, αλλά είναι ένα μέρος μιας προσπάθειας να απαντήσουμε πρέπει να ακολουθούμε και ε, τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Κομισιόν του κυρίου Γιούνκερ. Όπως ξέρετε, όπως ακούσατε, το μεταστευτικό είναι το βασικό πρόβλημα, η βασική, ο βασικός φάκελος που θα είναι συνέχεια μπροστά μας. Έχω μία μικρή ελπίδα ακούγοντας το άτυπο της ε, παρεμβάσεις των Υπουργών στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων ότι όλοι θέλουν, ε, συμφωνούν δηλαδή σε μια πιο ε, ενεργή στρατηγική έγινε η διάσκεψη στη Γενέβη προσπαθούμε να διοργανώσουμε και άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις ε, με δεσμευτικά συμπεράσματα, αλλά δεν είναι αυτή μία πολιτική που έχει, αναπτυ... έχει συντοπίσει όλα τα κράτη-μέλη. Έχω 13 κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει ορισμένε υποχρεώσει, έστω και μικρέ, και θέλουμε βεβαίω να βελτιώσουμε αυτή την κλίδα κατανομής. Αυτή η Frontex Βεβαίω θέλουμε κάθε πτυχή της Frontex να βελτιωθεί. Ίσως μπορεί η Frontex να συμμετάσχει στο μέλλον πιο ενεργά σε κοινέ σε κοινέ δράσεις και να κινητοποιήσει και συμπληρωματικούς πόρους, να δοθούν συμπληρωματικοί πόροι από άλλα κράτη-μέλη, από κράτη-μέλη τα οποία επισημούν ιδιαίτερα την ενίσχυση της Frontex. Αυτό το μήνυμα ακούμε και από την Ιταλική Προεδρία για το προφίλ των δράσεων που, θα, που επιθυμούν να υλοποιηθούν μέσω της Frontex μαζί με τη Mare Nostrum και τις συναφής δράσεις. πολλά από αυτά που λέμε ε, γίνονται και σε τρίτες χώρες. Η κυρία Γκόμες, η κυρία Γκυγιόμ έκανε μία ε, έκκληση ε, λέγοντας το πώς μπορούμε η αναπτυξιακή πολιτική, η πολιτική εξωτερικών υποθέσεων να συντονιστούν και να δουλέψουν καλύτερα μαζί. Είδαμε ότι και οι υπουργοί και άλλοι, οι συναρμόδιοι υπουργοί έχουν αναλάβει δεσμεύση ε, και για σας ως Επιτροπή θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Um, also a general point, but which is linked to the whole question of the common asylum system, but also και στο θέμα του ασύλου έχουμε μία τάση αυτή τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που δραστηριοποιούνται να λειτουργούν κάπως ε, ξεχωριστά, μεμονωμένα. Υπάρχουν κάποια στεγανά δηλαδή, ενώ η πολιτική αποφασίζεται στην, ε, στις Βρυξέλλες από εσάς, οι αποφάσεις λαμβάνονται εδώ, μετά προχωρούν προς τις υπηρεσίες ε, και τους φορείς όπου εκεί θα πρέπει να εφαρμοστούν και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οι φορείς συνεργάζονται μαζί μας. Ε, εγώ δεν λέω ότι δεν το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να συγκεράσουμε όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας με τον βέλτιστο τρόπο. Και θα πρέπει αυτό να το εξασφαλίσουμε ε, το ταχύτερο για να δουλεύουμε όλοι μαζί και συντονισμένα. Ε, πολλά θέματα εδώ έχω σημειώσει, στα οποία ε, σίγουρα επισημείτε συγκεκριμένε απαντήσεις. Uh, και τώρα δεν μπορώ βεβαίως ε, να τις αναφέρω όλες, ούτε κατά διάνοια να τις απαντήσω. Παραδείγματος χάρη αυτό που ακούγεται για μια ιδιωτική οργάνωση που θα αναλάβει διάσωση, τη διάσωση προσφύγων ή ε, αυτά, ούτε καν, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω αλλά σίγουρα χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να τα συζητήσω όλα αυτά. και ε, ε, το συντομότερο σε μια επόμενη συνεδρίαση θα προσφέρω περισσότερες απαντήσεις. Θα το, θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές, θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με τη συζήτηση αυτή Οπότε και τότε μπορείτε και εσείς ε, να έρθετε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί ετέθησαν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Νομίζω ότι έχετε σημειώσει πολύ διεξοδικά ε, όσα σας είπαν οι συνάδελφοί μου. Είμαι βέβαιος ότι με τα χαρά θα απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Οπότε απαντήστε σε αυτά τα ερωτήματα και εμείς οι συντονιστές θα τα συζητήσουμε και θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε κάποια άλλα συγκεκριμένα ε, βήματα για αυτή την ειδική ομάδα. Όποιος λοιπόν συνάδελφος ε, έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Μέχρι το Σεπτέμβριο ή το Σεπτέμβριο θα πάρει απάντηση συγκεκριμένη. Κύριο Σιρούτε, βεβαίω ε, με τα χαρά να το πράξω αυτό και διμερό με ορισμένου από του συναδέλφου σα θα μπορούσα να συζητήσω. Σίγουρα θα ήταν καλό να έχουμε μια σχέση εργασία, συνεργασία με όλου σα. Αν θέλετε, μπορώ και εκτός εθούσης να σας περιμένω τώρα ε, να συζητήσουμε, να δώσω απαντήσεις ε, σε όποιον το επιθυμεί. Και το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δώσω αναλυτικά τις απαντήσεις μου. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ιταλική Προεδρία και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Περνάμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είτε το πρωτόκολλο 36 της Συνθήκης Λισαβόνας προπαρασκευαστική εργασία εν ώψη της λήξης της μεταβατικής περίοδου την 1η Δεκεμβρίου 2014 επιλογή μη συμμετοχής opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου. Um, Όποιος θέλει να αποχωρήσει, ησύχως, αν μπορεί, παρακαλώ. Όσο αποχωρούν, όσοι αποχωρούν, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή εγώ. Όπως γνωρίζετε, υπήρχε ένα, ένα μεταβατικό, ένα προσωρινό πρωτόκολλο, το υπαρθμό 36 ε, για τη ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Είναι γνωστό αυτό στους Βρετανούς Συναδέλφου που άσκησαν την επιλογή τη μη συμμετοχή ίσω για άλλου συναδέλφου να μην είναι και τόσο γνωστό και βλέπω τεράστιο ενδιαφέρον από ορισμένου συναδέλφους. Περιμένω λοιπόν λίγο ε, οι Γάλλοι ναι, να αποχωρήσουν ησύχω. Εντάξει, ξέρω ότι είναι βρετανοβρετανικό το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε αυτό το πρωτόκολλο υπαρθμό 36 περιλάμβανε μία περίοδο μεταβατική διάρκειας 5 ετών. Θα συνεχίσω εγώ ε, να μιλάω, αν σας ενοχλεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και το σφυράκι μου. Πρώτη φορά το χρησιμοποιώ. Έλεγα λοιπόν το πρωτόκολλο 36 συμπεριλάμβανε μια μεταβατική περίοδο 5 ετών για να καθυστερήσει εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά μέτρα που είχαν να κάνουν με την αστυνομία και το ποινικό δίκαιο που είχαν εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και κυρίως ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Μετά το τελος μεταβατικης ματεβικής περίοδου 1η Δεκεμβρίου 2014, το άρθρο 10, εδάφιο 4 πρωτοκόλλο 36 των συνθήκων της Ένωσης δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο το αργότερο στην 31η 2014 αποφασίσει ε, εάν θα συμμετέχει ή όχι στα αστυνομικά μέτρα και μέτρα ποινικού δικαίου, τα οποία εγκρίθηκαν πριν την 1η Δεκεμβρίου 2009. Στο αποτέλεσμα όλα το μη λησβονοποιημένο, αν μπορώ να το πω, έξι ε, τέος ε, και εκτιμένο του τρίτου πυλώνα πάβει να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2014 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με επιστολή της 24ης Ιουλίου 2013, μόνιμος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει χρήση της επιλογής αυτής και να μην συμμετέχει στο τέος και εκτιμένο τρίτου πυλώνα. Με βάση το πρωτόκολλο 36 όμως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ε, να ενημερώσει το Συμβούλιο, του Ηνωμένου Βασίλειο, ότι επιθυμεί να συμμετέχει εκ νέου σε πράξεις οι οποίες έπαψαν να ισχύουν με βάση την απόφαση μη συμμετοχή. Στην νόμη του άρθρου 10, εδάφιο 5 του πρωτοκόλλου 36, ενημέρωσε επισήμω, μάλλον ανεπισήμω το Ηνωμένο Βασίλειο την του, για την πρόθεσή του να συμμετέχει ξανά στι 35 ε, μέσα αυτού του κεκτημένου σε 5 μέτρα Σέγγεν και 30 μη ε, Σέγγεν. Για να μην έχουμε νομικό επιχειρησιακό κενό, ε, προτείνει το νούμερο Βασίλειο ε, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014 να δοθεί έγκριση να μπορεί πλέον ε, να συμμετέχει σε αυτά τα 35 μέτρα το Συμβούλιο θα αποφασίσει με βάση τι συνθήκε για το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου ό,τι αφορά το κοινωνικό, ε, το κεκτημένο του Σέγγεν με ομοφωνία και έχει την ευθύνη η Κομισιόν να εξετάσει τα αιτήματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα μη Σέγγεν. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, αντιπροσωπεία και το Συμβούλιο τον Μάρτιο, τον προηγούμενο. Πρώτη ε, ανταλλαγή απόψε 10 Απριλίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. 16 Ιουνίου ο Γενικό Γραμματέα Επιτροπή έστειλε στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου ένα ανεπίσημο έγγραφο που διαβάστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών και περιλαμβάνει σύνοψη συζητήσεων, συνεχίζω τη συζήτηση και ολοκληρώνω. Πρέπει το Κοινοβούλιο ε, να δώσει την άποψή του για το σημαντικό αυτό θέμα και γι' αυτό θα έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και την Προεδρία. από την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα καλά, όλα καλά, μάλιστα. Έχουμε αλλαγές ε, στους ε, εκπροσώπους, δεν ξέρω ποιοι είναι, από την νομική υπηρεσία είναι ποιος. Ντάρτεν Τσουκ ή κάπως έτσι. Και από τη γάμα δέλτα Just της Κομισιόν είναι ο κύριος Στέλ Κυρία Σύπαλα είναι εδώ από την γάμα δελτα ΧΟΜ της Κομισιόν και δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Ίσως ε, ο εκπρόσωπος νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Καλά είπατε το όνομά μου. Όπως υπενθυμίσατε κι εσείς, δεύτερη, για δεύτερη φορά έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την κατάσταση ε, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 36. Γιατί αυτή τη δέσμευση έχουμε αναλάβει, δηλαδή να τηρούμε ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Την προηγούμενη φορά, 10 Απριλίου όπως είπατε, η Επιτροπή Ευρωπαϊκή εξήγησε ότι σε αυτό το πλαίσιο δύο πτυχές μας απασχολούν. Αφενός ε, ε, η λήξη, το τέλος μεταβατικής ε, περίοδου για τις ε, πράξεις του πρώην τρίτου πυλώνα, κάτι που ισχύουν για όλες τις χώρες Ένωσης και αφετέρου δυνάμει του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου 36 τη δυνατότητα μη συμμετοχή, το opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς οριστικοποιήσαμε τη χαρτογράφηση του σχετικού κεκτημένου που βρίσκεται και στο σχέδιο εγγράφου του Μαΐου είναι το επιχειρησιακό έγγραφο 2014-01-66 και εξετάζουμε τώρα κατά πόσον είναι πεπαλωμένες, απαρχαιωμένες ορισμένες νομικές πράξεις μπορούν λοιπόν να καταργηθούν και να ισχύει η επικαιροποιημένη νέα νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά το συνολικό ε, opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρετε ότι άσκησε το δικαίωμά του Ηνωμένου ε, μιας γενικής μη συμμετοχής, ε, ε, πέντε μέτρα συνολικά και άλλα 35, στα οποία θέλει να ξανασυμμετάσχει. Opt back in, σε αυτά θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δι, επι, διαλειτουργικότητα κτλ. Όλα αυτά ε, τα εξετάσαμε, το Συμβούλιο ό,τι αφορά το κεκτημένο Σέγγεν και η Κομισιόν ό,τι αφορά το σκέλος μη Σέγγεν. Η Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο κατέληξαν σε συνεννόηση ό,τι αφορά τεχνική ανάλυση των προτάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για να ξανασυμμετάσχει ε, στην, στο μη Σέγγεν κομμάτι μετά και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε ε, τα σχετικά. Βέβαια, επίσημη απόφαση μπορεί να ε, ληφθεί μόνο την 1η Δεκεμβρίου του 2014 Οπότε την ευθύνη για την ε, λήψη των αποφάσεων από πλευρά Επιτροπή θα την έχει το Σώμα των Επιτρόπων το καινούριο. Βέβαια, ήταν σημαντικό ήδη από τώρα να έχουμε πολιτική συνεννόηση, γιατί είναι σημαντικά ζητήματα αυτά και δεν θέλουμε να υπάρχει κανένα κενό την 1η Δεκεμβρίου. Ναι, μεν λοιπόν, όλε οι επίσημε αποφάσει εκκρεμούν, δεν θα ληφθούν τώρα, Έχουμε καταλήξει συνεννόηση και αυτό συμπεριλαμβάνεται και στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιο είναι το καθήκον της Κομισιόν ε, πολύ συγκεκριμένα ήταν να δούμε τις προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, που θέλει δηλαδή να ξανασυμμετέχει και θέλαμε να υπάρχει νομική ε, συνέπεια για να δούμε αν υπήρχαν επιχειρησιακά προβλήματα για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένες και όχι άλλες νομικές πράξεις. Το πρωτόκολλο 36 δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενική εξουσία να υπαγορεύσει το Ηνωμένο Βασιλείο σε ποιε πράξεις θα ξανασυμμετέχει συζητήσαμε και εξετάσαμε πιο διεξοδικά ορισμένες πράξεις, καταλήξαμε στο ότι τρία μέτρα εκτελεστικά ε, για κανονισμούς της Europol πρέπει να προσθεθούν, όπως και η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχθηκε την επιχειρηματολογία μας σχετικά. Κάποια άλλα ζητήματα επιλήθηκαν σε ό,τι αφορά τη λισαβονοποίηση, ε, όταν δηλαδή έχουν τροποποιηθεί κάποιε πράξει του τέο ε, τρίτου πυλώνα, έχουν καταργηθεί μετά την άρξη τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αφαιρούνται από τον κατάλογο ε, των πράξεων ε, του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου 36, άρα δεν υπόκεινται πια σε αυτή την ομαδική επιλογή μη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασίλειου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχθηκε επίση τα επιχειρήματα για τις αποφάσεις του δικτυου ΣΥΣ. SIS-2 δηλαδή το σύστημα πληροφοριών Schengen ε, που το συμβουλεύονται οι συνοριοφύλακες και η ε, αστυνομία. Άρα συμμετέχει ξανά σε αυτή την ε, συμφωνία. Σημαντικά βέβαια πολύ σημαντικά, αυτά τα ζητήματα για την επιβολή της νομοθεσίας, για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε να εξετάσει την πιθανή συμμετοχή του και σε μία δέσμη άλλων ε, τριών των αριθμό ε, πράξεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και την απόφαση ε, για την αναστολή και την προσωρινή κράτηση. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου για την υλοποίηση αυτών των τριών πράξεων πριν. Αυτά θα πρέπει να τα επιστρέψει εάν δεν συμμετέχει στο πριν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θα ε, συμμετέχει και στη μελέτη που θα εκπονήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, στη μελέτη αντικτύπου. Παρομοίως, αν αποφασίσει στα τέλη αυτή τη διαδικασία του Ηνωμένου Βασίλειου να μην ξανασυμμετέχει στο πριν, θα υποβάλει Κομισιόν ε, έκθεση που θα αναφέρει τις επιπτώσεις από την απόφαση αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ό,τι αφορά το probation, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει τις δεσμεύσεις οποίες ε, θα καταγραφούν στα πρακτικά του Συμβουλίου. Όλες αυτές τις συζητήσεις ε, τις παρουσίασαν στις 24 Ιουνίου στο σχετικό Συμβούλιο και προσπαθούμε και με το σκέλος του Σέγγεν να καταλήξουμε σε μια αντίστοιχη συνεννόηση. Για να παραμείνουμε εντό χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου και να έχουμε και μια ομαλή μετάβαση την 1η του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε ένα αντίστοιχο μνημόνιο συνεννόηση κατά κάποιο τρόπο να επιτευχθεί και με το Συμβούλιο. Αυτά και ολοκληρώνω εγώ τη δική μου παρουσίαση, ο πρόεδρος. Να ακούσουμε και την Προεδρία, αλλά να την παρακαλέσω την Προεδρία να είναι λίγο πιο σύντομη από τον προηγούμενο μιλητή, ή δυνατόν. Αν μπορείτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ναι, ναι, ναι, γιατί τα εξήγησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι η Ιταλική Προεδρία παίρνει τη σκητάλη από την Ελληνική Προεδρία, η οποία έκανε καταπληκτική δουλειά. Ήταν αφοσιωμένη, προσιλωμένη και εμβάθυνε πολύ σε αυτά τα θέματα όπως έκανε και η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα μέτρα Σέγγεν. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Είχαμε μια πρώτη ε, συζήτηση σε επίπεδο υπουργικό στο Συμβουλό Γενικών ε, Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία γνωρίζοντας ότι τα νομικά κενά πρέπει να τα αποφύγουμε την 1η Δεκεμβρίου του 2014. Και σίγουρα πρέπει να τηρήσουμε και το πνεύμα του πρωτοκόλου που ΕΕ θέλει να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει συνεργασία με το Ενωμένο Βασίλειο ε, όσο το δυνατόν ευρύτερη στα θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων. Αυτά είχα να πω. Είναι και νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να απαντήσει. Ε, σε ερωτήσεις, χωρίς να λέω ότι πρέπει να θέσετε ε, ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων ε, υποχρεούμε να σας το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, Δίας Ντεμέρα και Κέρκοπ είναι οι δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει μέχρι τώρα το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι. Δίας Ντεμέρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τη Μόνικα Χολμάγερ θέλω να ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως, διότι μου έδωσε εμένα το λόγο. Φίλεν Ντάνκ Μόνικα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε, διότι κατάλαβα πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο μας ε, μεταφέρατε σε όρθια αφορά το πρωτόκολλο 36 και τη θέση του Ηνωμένου Βασίλειου. Βέβαια δυσκολεύτηκα πιο πολύ να καταλάβω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το Συμβούλιο το κατάλαβα, τέλος πάντων. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, ευχαριστώ όλους όσους έχουν λάβει μέχρι τώρα το λόγο για να ε, χύσουν φως ε, σε αυτή την υπόθεση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας ε, πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα ποινικού δικαίου. Καταλαβαίνω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όπως είναι φυσικό, ασκεί τα δικαιώματα ε, ε, που του, που του έχουν εκφορήσει οι συνθήκες. Ε. Αλλά εμείς θα θέλαμε να μην αποχωρήσει από το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έστω εν μέρη. Είναι νησιωτική περιοχή μένα, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό κράτος. Θέλει, μπορεί, μάλλον δεν θέλει, δεν μπορεί να συμμετέχει συνολικά στο χώρο της ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας ε, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει να κάνει, αλλά θα ήθελα για τα πολύ ευαίσθητα λεπτά αυτά ζητήματα να ε, συμμετέχει. Δηλαδή ασφάλεια, ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας, ε, το ΠΡΙΜ, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, δραστηριότητες ορισμένων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, φορέων, όπως είναι η Europol. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά ε, και εκεί πρέπει να αναζητήσουμε την ε, μέγιστη δυνατή συνεργασία και την απαιτούμενη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνικών, ε, κοινοτικών συγγνώμη, εταίρων. Πρέπει να αποφύγουμε, κύριε Πρόεδρε, και το λέω ιδίως στον αγαπητό φίλο Κίρκοπ, πρέπει να αποφύγουμε την επιλεκτική συμμετοχή για μια ακόμη φορά σε ορισμένους από τους ε, το 35 μέτρα κτλ. Γιατί πραγματικά επηρεάζεται η εφαρμογή ε, των συνιστοσών του κοινοτικού και εκτιμένου στον τομέα της ασφάλισης αφαιρές δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνεκτικότητα των συνιστοσών αυτών. Πρέπει να υπάρχει σαφής βούληση συνεργασίας με σεβασμό στα κριτήρια του πρωτοκόλου 36. Δηλαδή, απλούστευση, αναζήτηση της μέγιστης δυνατής συνεργασίας στον τομέα αυτό, διευκόλυνση της επιχειρησιακής ε, λειτουργίας όλου του συστήματος και εξασφάλιση της ε, συνέπειας και συνεκτικότητας. Για να μην ε, φλιαρίσω άλλο, κύριε Πρόεδρε, διότι αφορά το εκτός Σέγγεν και Σέγγεν, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, Απλά απευθύνω αυτή την έκκληση στους Βρετανούς συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στεμέρα. Χαίρομαι που τα είπατε αυτά γιατί έχετε δουλέψει σε αυτούς τους τομείς και αυτή ε, αυτοί οι τομείς είναι ε, αντικείμενο αυτής της ε, επιλογής συμμετοχής ή μη συμμετοχής. Ε, υπάρχουν και άλλοι ε, ομιλητές. Ε, πρόκειται όμως πριν πάρει το λόγο ο κύριος Κέρκοφ να πω ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής ελπίζω να πετύχει αυτή η επιθυμία επιστροφής, συμμετοχής. Θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι ελπίζουμε να πετύχει αυτό. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε διάλογο φυσικά. Ο κύριος Κέρκοφ. Θέλετε ίσως να επισημάνετε κάποια από αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι ήμουν πολύ ευτυχής επί πολλά χρόνια που μου δόθηκε δυνατότητα μεταξύ των άλλων να συνεργαστώ στενά με τον κύριο Δίας Ντεμέρα για εξαιρετικά μεγάλη σημασία θέματα για την Ευρώπη στον τομέα της ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ε, αρχών επιβολής του νόμου που ασχολούνται με εγκληματίες και τρομοκράτες, θέματα για τα οποία και εκείνος και εγώ έχουμε άμεση εμπειρία. Στο επίπεδο λοιπόν αυτό είναι σημαντικό να το θέσω. Δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και όλοι οι άλλοι παριστάμενοι κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ε, κοινοβουλευτικό ζήτημα εδώ. Είναι θέμα ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Η αυτοί που είναι καλύτεροι από εμά στις εθνικές κυβερνήσεις και που έχουν σχέση με τις συνθήκες και τους συγκεκριμένους τομείς του πρωτοκόλλου αυτού. Είμαι από τους δικηγόρους που ασχολούνται με το, το θέμα του τρίτου πυλώνα και πριν από το 2009 ήταν απόλυτα σαφές σε μένα ότι υπήρχαν τομείς που υπήρχε εθνική αρμοδιότητα σε πολλά πράγματα. Αυτό έληξε με τον τρίτο πυλώνα μετά το 2009. Ε, καταστράφηκε ένας πυλώνας, παρά τα αυτά ε, ε, ε, αντιμετωπίστηκε εν πάση περιπτώσει με, με διαφορετικό τρόπο. Και ε, θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι από το 2009 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια πολύ θετική ε, στάση επιλογής συμμετοχής σε αυτό του τομείς που συζητάμε εδώ. Μιλάμε τώρα για την περίοδο πριν από το 2009, ένας, μια σειρά θεμάτων όπου υπήρχε δυνατότητα να επιλέξουμε να μην συμμετέχουμε. Χαίρομαι όμως πολύ που μοιάζει να, ότι προχωράμε πολύ καλά και είναι στο, στο συμφέρον όλων μας, κυρίως στον τομέα της Europol, κάπως με, με κάποια μεταρρύθμιση, μια σαφήνεια όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ε, μια συνεργασία που μου φαίνεται εφικτή. Πιστεύω ότι υπάρχουν ανάμεσα στα πολλά πάνω από 100 ζητήματα ένας αριθμός που θα έλεγα, παρότι και εγώ συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις, θα, εγώ θα έλεγα ότι έχουν ξεπεραστεί ή είναι περιτά και το γνωρίζουν και άλλοι αυτό. Και αν αυτή η διαδικασία έχει παράξει κάτι που είναι να μας κάνει να κοιτάξουμε σε άλλους τομείς όπου υπάρχουν περιττή κανονισμοί και περιττές διατάξεις και αν μπορούμε αυτά να τα διαχωρίσουμε, κατά τη γνώμη μου το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό είναι να προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους, στους λαούς της Ευρώπης για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παραπροϊόν αν θέλετε, αλλά είναι θετικό. Επίσης, στην όλη αυτή διαδικασία Χάρηκα πολύ που άκουσα τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία και σαφώς ε, στη συζήτηση που είχα στο Λονδίνο υπήρξε πολύ θετική ε, στάση από τους αρμόδιους υπουργούς μας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, τη σημασία και την επιτυχία, τις επιτυχίες των διαπραγματεύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει πλήρως ε, συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν τα σοβαρά δικήματα και άλλους τομείς όπου οι δυνατότητες επιστροφής μας δίνουν τώρα αυτή τη δυνατότητα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσουν στο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Um, very nice. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ε, βλέπω ότι ε, ε, υπάρχει χειραψία εδώ, είναι καλό. Θέλω να πω ε, στα μέλη της Επιτροπής γιατί έχει μπει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Γιατί εάν επιτύχει αυτή η επιλογή συμμετοχής όπως ελπίζουμε, Θέλω να διορθώσω ότι έχει νομοθετική επίπτωση. Η μη εφαρμογή έχει ε, νομοθετική επίπτωση και οικονομική επίπτωση. Το Κοινοβούλιο ε, έχει ένα συμφέρον, εδώ, έστω και περιορισμένο πρέπει πάντοτε το πρωτόκολλο 36 να είναι στην ημερήσια διάταξη. Το, θέλω να σας το εξηγήσω αυτό. Μην φανταστείτε ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί, αλλά υπάρχουν καθαρά κοινοβουλευτικοί λόγοι, νομοθετικοί λόγοι. Τώρα, ε, Σόφη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως Θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Δεν μου αρέσει η επιλογή συμμετοχής και η κατεπιλογή ε, συμμετοχή μια χώρα που δεν είναι στο Σέγγεν, που επιλέγει να μην συμμετέχει στην δικαστική και πολιτική συνεργασία, που αν δεν κάνω λάθος δεν έχει προσυπογράψει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και που δεν συνεργάζεται σε πολλούς άλλους τομείς. Τώρα έχει τη δυνατότητα επιλογής ε, για να επιστρέψει. Σας παρακαλώ, όπως ε, ε, πολύ πιο διπλωματικά είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα και οι περισσότεροι άλλωστε το είπαν πιο διπλωματικά από ότι εγώ. Ανησυχώ για την ε, συνοχή της, ε, των πολιτικών μας αλλά και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είπατε ότι αυτό έχει νομοθετική επίπτωση αλλά επηρεάζει και τον τρόπο της δουλειάς μας εδώ. Διότι πώς λειτουργούμε μεταξύ συναδέλφων αν οι συνάδελφοι αποφασίζουν επί κάποιου θέματος ότι η χώρα τους δεν συμμετέχει. Είχαμε και στο παρελθόν, στην προηγούμενη θητεία, στην Επιτροπή Οίκων, την κατάσταση όπου προτάθηκε, αλλά ευτυχώς δεν ε, εγκρίθηκε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να δημιουργηθεί μια χωριστή επιτροπή εντός του Κοινοβουλίου που θα αποτελείται από μέλη των χωρών ε, ε, της Ευρωζώνης. Θα κόψουμε και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και στην πράξη είσαι αστυνομικός που θα έχει στο γραφείο σου έναν κατάλογο των τομέων στους οποίους συνεργαζόμαστε και τους τομέων στους οποίους δεν συνεργαζόμαστε. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος στην πράξη δεν θα ξέρει πού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αρμόδιο και πού δεν είναι. Που ε, ε, ισχύουν οι κανόνες των δημιουργικών δικαιωμάτων και που δεν ισχύουν. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση, καθόλου δεν μου αρέσει. Συμφωνώ, δεν μπορώ να αλλάξω μόνη μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να πω ότι με, δεν με ικανοποιεί καθόλου και θα ήθελα να υπήρχε ένα μπλοκ, ένα ε, για την επιλογή επιστροφής. Ο κύριος Κέρκοφ είπε θέλουμε να συμμετάσχουμε πλήρως. Λοιπόν, να συμμετέχετε πλήρως σε όλες τις πολιτικές. Αν αντιμετωπίζουμε την αντιμετώπιση του εγκλήματος της τρομοκρατίας και των κακών με σοβαρότητα, αυτοί διατρακινούνται στα σύνορα με ελευθερία. Δεν κάνουν ε, ούτε επιλογή να μπουν, ούτε επιλογή να βγουν. Δεν λένε ότι θα κάνουμε κάποια αδικήματα σε κάποιες χώρες και κάποια άλλα αδικήματα σε άλλες χώρες. Βεβαίως και δεν το σκέφτονται αυτό. Λοιπόν, τελευταία παρατήρηση. Ο Τιμισή είπε ότι ίσως θα πρέπει με την ευκαιρία αυτή να απαλλαγούμε από τις ε, πλεονάζουσες διατάξεις. Αυτό με κάνει να μιλάω με κινησμό, γιατί αν υπήρχε μία χώρα, μία χώρα που ζητά όλο και περισσότερα μέτρα στον τομέα της ε, ε, ασφάλειας και της διοξής, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Κυριάρχησε αυτό όλες τις συζητήσεις και έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά... Είτε παίζεις με τους όρους μας είτε δεν παίζεις. Έτσι λοιπόν, σας ζητώ να επιλέξετε την επιστροφή σας στο χώρο της ε, συνεργασίας ε, δικαιοσύνης και αστυνομίας και να συνεργαστούμε στο 100% τον επόμενο, το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Uh, you got that, <laughs> did you, Timothy? okay, thank you very much, Sophie. Λοιπόν, ευχαριστώ Σοφία. Όπως είπε και ο κύριος Δίας πιο διπλωματικά είπε το ίδιο πράγμα με σας. Δεν ξέρω τι από τα δύο προτιμώ. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Πρέπει το θέμα να τεθεί, να τεθεί για τους λόγους που ανέφερα. Ας προχωρήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε για την ανοχή και την αντοχή σας. Περνάμε στο επόμενο θέμα υπαριθμών 8 προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Είναι ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Ο Γιάνν. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα δώσω το λόγο στο Γιάννη. Έχουμε το πακέτο της μεταρρύθμισης ε, της προστασίας των δεδομένων, η οποία υπερψηφίστηκε στις 12 Μαρτίου ε, με συντριπτική πλειοψηφία. Τα λέω αυτά για τα νέα μέλη. Ο κύριος Άλμπρεχτ ήταν ο εισηγητής και θα μας κάνει μια παρουσίαση για το πού βρίσκεται το θέμα. Θα δώσω το λόγο και σε αυτόν και στους κοιόδης εισηγητές που παρευρίσκονται. Οι σκιώδεις εισηγητές είναι ο κύριος Βος, ο κύριος Κάρκοφ, η Κορνίλια Έρνστ, όλοι παρίστατες. Γιάν, σε παρακαλώ, έχεις το λόγο. Τιμωθεί θα μείνεις για το, να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ε, κουράστηκες. Εντάξει, εντάξει. Έχεις άλλη συνεδρίαση, εντάξει. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω διάλογο με ένα μέλο που αναχωρεί. Ε, λοιπόν, συγγνώμη. Γιαν έχεις το λόγο. Thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω καταρχάς το προηγούμενο ιστορικό ε, για όλη αυτή την ιστορία της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσωπικού χαρακτήρα και για την τρέχουσα κατάσταση. Το θέμα ξεκίνησε όταν ζητήσαμε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την οδηγία 95-46 και η οδηγία αυτή τότε ζητούσε μία αναθεώρηση για να δημιουργήσουμε ένα υψηλότερο πρότυπο για την ε, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που να σέβεται τα δικαιώματα των ε, φυσικών προσώπων, ε, στο διαδίκτυο, να ενισχυθεί η διαφάνεια και για να εδραιωθεί ένας μόνιμος ε, μηχανισμός ε, ε, υλοποίησης αυτών των διατάξεων. Υπήρχαν βεβαίως μεγάλες διαφορές μεταξύ των τομέων τους οποίους κάλυπτε αυτή η νομοθετική πράξη. Το, η πρόταση λοιπόν το 2012 ήταν να δημιουργηθεί ένας κανονισμός που θα αντικαθιστούσε την οδηγία 9546. Αλλά θα ε, ε, αποκλείονταν από το πεδίο εφαρμογής ε, η, η συλλογή πληροφοριών και συναφής τομείς. Από τον Ιανουάριο του 12 λοιπόν δουλεύουμε πάνω σε δύο φακέλους την οδηγία και τον νέο κανονισμό εκ παραλίλου και τα συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Εγώ ήμουν εισηγητής για τον κανονισμό και ο κύριος Δρούτσας ήταν ο αρμόδιος εισηγητής για την οδηγία. Και τελικά καταλήξαμε σε αυτή την Επιτροπή μας ε, πέρσι τον Οκτώβριο σε μια απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία επί τη βάση πολλών τροπολογιών που υποβλήθηκαν και μετά από πολλούς ε, διαπραγματευτικούς γύρους, συνεδριάσεις, συζητήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες ε, αποφασίσαμε στο να ανοίξουν οι διαβουλεύσεις ε, στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και αυτός ο άτυπος ε, τριμερής διάλογος, αυτή η διαβούλευση δεν άρχισε ποτέ διότι το ε, Συμβούλιο δεν κατέληξε σε γενική προσέγγιση πριν από τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου. Οπότε χρησιμοποιήσαμε το, τη δεύτερη εναλλακτική λύση ε, να το συζητήσουμε στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Από το Μάρτιο λοιπόν φέτος εμείς ως Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε την θέση την οποία η Επιτροπή επεξεργάστηκε πάνω σε αυτά τα δύο ντοσία και περιμένουμε τώρα από το Συμβούλιο να μας ανακοινώσει τη θέση του. Είναι περίπου δυόμιση χρόνια, δεν έχουμε ακόμα τη θέση του Συμβουλίου. Είναι μία μακρά διαδικασία, δεν λέω, μες στο Συμβούλιο αλλά πρέπει και να προσθέσω ότι αυτή είναι μια ατυχής, ένα ατυχό, ατυχές παράδειγμα, μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ε, δεν μπορούμε εμείς ε, να τους πούμε με μετήρησιμο θα δουλέψουν, αλλά πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι, εν πάση περιπτώσει, ας καταβάλουν προσπάθειες να εργαστούν λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσει να αρχίσει ο τριμερής διάλογος και να καταλήξουμε ποιες είναι οι κοινέ θέσεις και ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει ακόμα να διευθετηθούν. Το τελευταίο άτυπο συμβούλιο έγινε πριν από μερικές εβδομάδες όπου παρουσιάστηκε το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της Προεδρίας και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα προσπαθήσουν να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε μια γενική προσέγγιση το οποίο ελπίζω να σημαίνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Και η επόμενη ευκαιρία για συζήτηση με το Συμβούλιο τον Οκτώβριο και θα δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και τι θα αποφασίσουν εκεί αν μπορέσουν τελικά να διατυπώσουν μια γενική προσέγγιση ε, είτε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου είτε αμέσως μετά. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, επί της ουσίας, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία επανέρχονται στο Συμβούλιο ε, φαίνεται ότι έχουν λυθεί με τη θέση και τους συμβασμούς που έχουμε επιτύχει και όλο και περισσότερο το Συμβούλιο το αναγνωρίζει αυτό ότι έχουμε κάνει πολλές φορές τις ίδιες συζητήσεις για τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το δημόσιο τομέα, ε, διαφορετικές ε, ρυθμίσεις για την μόνιμη εφαρμογή αυτή της νομικής πράξης στην επεξεργασία δεδομένων ε, ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική αγορά όπου ε, αυτή θα είναι και το κύριο πεδίο υλοποίησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ε, υλοποίηση με συνέπεια, συνεπής, έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μία ερμηνεία και όχι 28 συνεχώς ε, εξελισσόμενα και ε, μετατρεπόμενα, ε, μετατρεπόμενες νομικές πράξεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ενιαία και συνεπή εφαρμογή. Πιστεύω λοιπόν ότι το Συμβούλιο ε, θα μπορούσε ανετότατα να δει την δουλειά μας όλη αυτή και να την υιοθετήσει ως έχει, να την κοπιάρει θα έλεγα. Ε, εν πάση περιπτώσει θέλουμε την ε, απάντησή του το ταχύτερο. Αυτή είναι η θέση μας ε, του νέου κοινοβουλίου και καταλήγοντας θέλω να πω ότι ε, και είμαι πολύ σαφής ότι αυτή η νομοθετική πράξη ήταν μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για αυτό το σώμα και θα θέλουμε να δημιουργήσουμε την ίδια διαδικασία και άλλες νομοθετικές πράξεις για να μπορέσουν να υπερψηφιστούν δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός με άλλες αγορές παγκοσμίες και με άλλες ε, δικαιοδοσίες ε, που ακόμα έχουμε εσωτερικό δικαιοδοτικό ανταγωνισμό μέσα στη δική μας επικράτεια. Αυτό το τονίσαμε πολλές φορές ε, πέρσι με όλα τα προβλήματα της παρακολούθησης και στο ψήφισμά μας το τονίζουμε αυτό, του Κλόντ του που ήταν εισηγητής. Επαναλάβαμε όλα αυτά τα σημεία και ε, επίσης επιμείναμε στην ε, αναστολή της απόφασης These περί για να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη προστασία των φυσικών προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομος. Και όσοι δεν ξέρουν τα, θέματα αυτά του κανονισμού και της οδηγίας είναι πολύ κρίσιμα. Και θέλω ε, να είναι όλοι ενήμεροι και οι συγητές και οι, και οι σκιώδεις συγητές. Γι' αυτό θα ήθελα να τους δώσω το λόγο. Έχουμε μέχρι τις ε, μισή καιρό. Λοιπόν, καταρχάς, Κομισιόν, Προεδρία, αλλά παρακαλώ τηλεγραφικά. Καταρχάς, Προεδρία. 1,5 λεπτό ή δυνατόν, γιατί έχω και ένα μακρύ κατάλογο μελών που θέλουν να μιλήσουν. Μετά από τις 5.30 έχουμε την συνεδρία κυκλισμένων των θυρών. Λοιπόν, από πλευράς Προεδρίας, ο κύριος Ντεματίας από πλευράς Ταλικής Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ε, με μεγάλη χαρά, χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και πιστεύω ότι ε, στη νέα τι θα προχωρήσουν ικανοποιητικά και ο κανονισμός και η οδηγία για την προστασία δεδομένων. Είναι σαφής ε, προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας, όπως είπε ο Υπουργό το πρωί γιατί ε, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ε, Ευρωπαίων πολιτών και για τις εταιρείε και για τους οικονομικούς τομείς. Πρέπει κανείς λοιπόν να δικαίως οι πολίτες μας αναμένουν από εμά τη δημιουργία ενός ε, σταθερού ισχυρού νομικού πλαισίου. Στο Συμβούλιο γνωρίζουν σαφώς ε, ότι δυόμιση χρόνια συζήτηση είναι μια πολύ μακρά περίοδος και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι διαβουλεύσεις στην οδηγία ε, που προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Δεδομένου ότι δίνει μεγαλύτερο εύρος διαχείρισης στα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Συμβουλίου, πρέπει να κάνουμε υπομονή, που να δούμε τι θα αποφασίσουν στα τεχνικά θέματα έχουμε ουσιώδεις συμβολές από τα κράτη-μέλη. Δεν έχει χαθεί ούτε μία μέρα διαπραγματεύσεων. Στην ε, Προεδρία πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουμε την επιτυχία ε, των ενεργειών της ελληνικής προεδρίας και των προηγουμένων ε, προεδριών και θα συγκεράσουμε όλες τις προηγούμενες εργασίες σε μια συμβιβαστική πρόταση την οποία πιστεύω ότι θα, μπορεί, θα γίνει αποδεκτή υπάρχουν ακόμα εκκρεμή θέματα, σοβαρά κρεμή θέματα. Ε, έχουμε ε, τις απόψεις ε, κρατών μελών που έχουν συγκεράσει διαφορές απόψεων μεταξύ συναρμοδίων φορέων και υπουργείων ε, πολλά σημαντικά πράγματα αποφασίστηκαν στην ελληνική προεδρία παραδείγματο χάρη στις, ε, στις διεθνείς, ε, στη διεθνή πτυχή των μεταφορών και μετά, μετάδοση μάλλον στοιχείων και δεν θα ήθελα να προτείνω μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Ε, αν, ε, αυτή τη στιγμή σας πω ότι θα είναι Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Το Συμβούλιο ε, λειτουργεί ικανοποιητικά. Η τελική Προεδρία θα υποστηρίξει τι του Συμβουλίου με όλες τις δυνάμεις και θα συνεργαστούμε όπως πάντα με το Συμβούλιο και θα σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε το ταχύτερο να αρχίσουμε διαβουλεύσεις με τους συνομοθέτες. Σας ευχαριστώ. Λέτε δεν θέλετε να μας δώσετε ημερομηνία. Αλλά εν είδη συμπεράσματος ε, λέτε κάποια πράγματα. Πότε θα ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Δεν μας δίνετε ημερομηνία και μας ε, λέτε περίπου πώς θα καταλήξουν αυτά. Ε, δεν έχουμε καμία αίσθηση για το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι. Φανταζόμουν ότι θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένος στο 1,5 αυτό λεπτό. Απάντησα, ακούστε, είναι δύσκολο κύριε Πρόεδρε, γιατί εξαρτάται από την εντολή που θα μας δώσουν τα κράτη-μέλη. Στο Συμβούλιο του Ιουνίου έδειξαν τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι διατεθειμένα να δώσουν εντολή σε καμία Προεδρία, ώστε ένα μέρος του κανονισμού να τεθεί σε διαπραγμάτευση προτού έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για ένα συνολικό εργαλείο ή μέσο. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να έχουμε αυτό το γενικό πλαίσιο. Να είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα ξεκάθαρο. Από τη δική μας πλευρά δεν είναι και πολύ ε, χρήσιμο να σας ανακοινώσουμε μια ημερομηνία μόνο και μόνο για να σας δώσουμε μια ημερομηνία. Εμείς εργαζόμαστε ώστε το συντομότερο δυνατό να έχουμε κάποια πρόοδο. Το τέλος του έτους είναι ρεαλιστική ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ, λάβαμε το μήνυμα. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν, παρακαλώντας τον εκπρόσωπο να είναι σύντομος. Σεστακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Κομισιόν λίγα πράγματα θέλει να πει από τότε που έγινε η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο το Μάρτιο ε, διαπιστώσαμε μία αλλαγή στη δυναμική των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και μεγαλύτερη προθυμία να, γίνει, ε, ε, να ολοκληρωθεί το θέμα γρήγορα. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στο Κοινοβούλιο που έκανε αναπόφευκτη αυτή την μεταρρύθμιση. Αισθανόμαστε ότι έχει δοθεί μία όθηση η οποία συνεχίστηκε και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Ε, ήταν ε, επιτυχημένο το Συμβούλιο του Ιουνίου πέρα από την ε, γενική προσέγγιση που επετεύχθη από την ελληνική προεδρία. Έγινε καλή συζήτηση για τον δημόσιο τομέα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης όπου έγινε σαφές ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών ενδιαφέρονται ο δημόσιος τομέας να παραμείνει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Τώρα ο ρόλος της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει την Προεδρία να δουλέψει το ταχύτερο δυνατό για να κλείσει τα θέματα ένα-ένα ώστε να δουλέψει αποτελεσματικά στο θέμα αυτό μετά το άτυπο, να κλείσει το θέμα του ε, one-stop shop και να διατηρηθεί η προσέγγιση κινδύνου που ε, προέβαλε η Ιρλανδική Προεδρία. Έτσι νομίζω ότι πρέπει αυτό να γίνει μέχρι το Δεκέμβριο. Επίσης είναι πιεστικό, πιέζει να διατηρηθεί το πακέτο. Νομίζω ότι αυτό σκοπεύει να κάνει και η Προεδρία ώστε ο, ο κανονισμός και η οδηγία να προχωρήσουν από κοινού. Μιλήσαμε για ημερομηνίε. Η πιο σημαντική ημερομηνία είναι αυτή που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μέχρι τότε που πρέπει να, ε, πρέπει έχει κλείσει ο φάκελος ε, μέχρι το 2015 και είναι μια ημερομηνία που πλησιάζει και πρέπει να την τηρήσουμε. Ναι, το 2015 πλησιάζει, επ' αυτού συμφωνούμε. Κάθε μέρα πλησιάζει και περισσότερο. Ε, εδώ γίνονται φιλοσοφικές συζητήσεις όπως βλέπετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε κατευθείαν στους σκιώδεις, στους συντονιστές. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα-δυο λεπτά για να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν, για να καταλάβουμε όλοι προς τα που κινούμαστε. Καταρχήν, ο κύριος Βος για τους Σκιώδης. Ευχαριστώ. Ε, όπως είπε και ο Γιάνν Άλμπρεχτ, Έχω το αίσθημα ότι όσο περισσότερο περιμένουμε στην Ευρώπη, τόσο περισσότερο θα βρισκόμαστε σε οπισθοχώρηση. Και βεβαίως, αφενός πρέπει να αποτανθούμε στην Κομισιόν η οποία θα πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες της, τις νέες θέσεις κλπ. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να αποταθούμε και στην νέα Ιταλική Προεδρία. Μήπως ε, Φίλιπ μπορείς ε, να πεις αν έχεις και την άποψη ας πούμε του, του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών, έχεις ακούσει τίποτα. Εγώ έχω το αίσθημα ότι αυτά τα, ε, αυτή η νομοθετική προστασία στοιχείων μπορεί να εμπλέξει και τον, τριμερό, τον τριμερή διάλογο πάλι σε μακρές συζητήσει. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα προχωρήσει γρήγορα. Το πρόβλημα που έχει το Συμβούλιο ίσως έγκυται στο ότι είναι κανονισμός και πρέπει να περάσει από όλους. Αλλά η ανάγκη να προχωρήσουμε είναι εμφανέστατη δεν πρόκειται μόνο για τις δημόσιες υπηρεσίες ή για το one-stop shop. Σε αυτά ίσως βρεθούν λύσεις, αλλά πρόκειται για όλο το φάσμα. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε πρώτα το πρόβλημα σε, ρεαλιστικό επίπεδο να έχουμε και την γνωμοδότηση του νομικού, της νομικής υπηρεσίας για να είμαστε σίγουροι ότι ένα τέτοιο άνοιγμα είναι και νομικά συμβατό. Ευχαριστώ. Ο, ποιος είναι ο καινούριος σκιώδης εισηγητής? Ε, ευχαριστώ. Σήμερα έλαβα ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσω τη δουλειά που έκανε ο κύριος Δρούτσας ως εισηγητής και όδης εισηγητής της οδηγίας. Ελπίζουμε, ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και είναι σημαντικό να διατηρηθεί η προσέγγιση συνολική πακέτο γιατί είναι ανόητο να υπάρχει η αντιμετώπιση της οδηγίας η οποία δεν θα έχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ζούμε σε μια εποχή ε, που είμαστε σε ψηφιακό ε, αυτοκινητόδρομο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε κάθε χώρα τα πράγματα να είναι ε, τα ίδια. Είναι πολύ καλό που η Ιταλική Προεδρία σχεδόν υποσχέθηκε ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν ομαλά όσον αφορά τον κανονισμό. Έχω αρχίσει να φοβάμαι όμως το σκέλος οδηγία. Ελπίζω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το πακέτο να προχωρήσει και ε, είναι πολύ σημαντικό για το TTIP και για την ψηφιακή κοινή αγορά υπάρχει ένα περιβάλλον ε, στο οποίο και τα δύο μπορούν να προχωρήσουν από κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλντε, ε, Σκιώδη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Δεν έχουμε πολλά να πούμε από αυτού τώρα. Όσον αφορά το θέμα του χρόνου, αν ήμουν κοινική, ενώ δεν είμαι, θα επιθυμούσα να καθυστερήσει το Συμβούλιο γιατί όσο καθυστερούν τόσο περισσότερη νομολογία θα έχει παραχθεί που θα ενισχύει την άποψη του Κοινοβουλίου και όχι του Συμβουλίου. Δεν μπορώ να προκαταλάβω φυσικά την θέση του Συμβουλίου, αλλά Ακόμα δεν έχω δει μια νομοθετική πρόταση όπου πήρε μια θέση το Κοινοβούλιο η οποία να βελτιώθηκε και να ενισχύθηκε από το Συμβούλιο. Κυρίως συνήθως την αποδυναμώνουν. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Η θέση του Κοινοβουλίου ήδη αποτελεί συμβιβασμό. Εκτός και θέλουν να την ενισχύσουν. Ευπρόσδεκτο αυτό από το Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συζητάνε επί τόσο μεγάλο διάστημα. Και εκτός αν θέλουν την αποδυναμώσουν την περαιτέρω. Και παραδέχομαι ότι παρότι συμφωνώ, συμφωνώ με τον Άλμπρεχτ, ε, ε, συμφώνησα με το συμβιβασμό του Κοινοβουλίου, αλλά απρόθυμα γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στο επίπεδο προστασίας. Υπάρχουν σημαντικά ερωτηματικά. Άρα το αν το Συμβούλιο θέλει να την αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο, δεν πιστεύω ότι μπορώ τελικά να την υπερψηφίσω. Πρέπει να κινηθώ προς τη θέση του Κοινοβουλίου και όχι να απομακρυνθούμε ακόμη περισσότερο από αυτή. Οπότε συνιστώ στο Συμβούλιο να κινηθεί σβέλτα και να προσεγγίσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κορνίλια. Λοιπόν, αυτή είναι ένας μακρύς δρόμος ε, τον οποίο ήδη έχουμε διανύσει εδώ και δυόμιση χρόνια, ίσως και περισσότερο όπως ελέγχθη. Ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε ως κοινοβούλιο να πούμε εμείς αρκετά κάναμε. Τώρα το μαύρο πρόβατο είναι το Συμβούλιο, είναι σκάνδαλο ότι δεν υπάρχει καν μία ημερομηνία κίνησης ε, του τριμερούς διαλόγου αποτελεί ένιγμα όλη αυτή η τακτική. Πιστεύω ότι είναι τακτική καθυστέρησης και είναι αντι... απογοητευτικό αυτά τα οποία ακούσαμε από το Συμβούλιο και οι απαντήσεις ήταν ε, τουλάχιστον κανένα ψήμου, κρυπτογραφημένες. Ε, ε, τίποτα συγκεκριμένο δεν ακούσαμε ότι θα υπάρξει σαφής κανονισμός και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Για την TTIP ελέγξει ότι δεν χρειάζεται ενσωμάτωση ε, των δεδομένων, προστασίας δεδομένων, διότι η TTIP θα σεβαστεί όλη την ε, νομοθεσία, την ευρωπαϊκή κλπ. ως πακέτο. Το ίδιο ακούσαμε και για το NSA, ότι ε, και, αυτό καλά να πάθουμε, γιατί για αυτό το πακέτο προστασίας δεδομένων το οποίο εξεργαζόμαστε τόσα χρόνια και με τέτοιες καθυστερήσεις που τελικά έχουμε χάσει τον έλεγχο και τα πράγματα έχουν τελείως χαλαρώσει, δηλαδή τα θέματα της προστασίας. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε μία συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης του τριμερού διαλόγου και όχι περαιτέρω καθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Κορνηλία. Άλλος επιθυμεί το λόγο παρακαλώ. Ο Τζόζεφ, Γιώζεφ είναι ο επόμενος. Δεν, δεν, δεν είμαι προκατηλημένος εναντίον της δική μου ομάδας, αλλά είναι η Μπριγκίτα Α, η θέλει. Λείπουν οι συντονιστές, οπότε τέλος πάντων η κυρία Ζίπελ παίρνει το λόγο. Μη δώσει σε άλλου το χρόνο που δικαιούμαι, λέει η κυρία Ζίπελ. Ωραία, ακούω τα λόγια, αλλά δεν βλέπω τη βούληση, τη θέληση. Όλοι λένε ότι το Συμβούλιο χρειάζεται χρόνο επειδή πρόκειται περί κανονισμού. Μάλιστα, και πρέπει να εργαστούμε με πολύ προσοχή. Μα συγγνώμη, δεν έχουμε πια καιρό και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο το Συμβούλιο εάν δεν είχε χάσει ατελείωτες εβδομάδες κλαψουρίζοντας ότι «Ω, μα δεν θέλουμε, δεν θέλουμε κανονισμό». Μα αυτό είναι ακριβώς η ουσία. Το Συμβούλιο δεν θέλει τον κανονισμό. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν καταλάβει ότι ο χρησμός αυτός είναι απέτηση, διότι χρειαζόμαστε ενιαία πρόταση για την επεξεργασία των δεδομένων, των στοιχείων. Δεν έχουμε πια καιρό, δεν έχουμε πια καιρό. Η ψηφιοποίηση όλων των τομέων ε, προχωράει με ακατάσχετους ρυθμούς και δεν θα περιμένει τις δικές μας αποφάσεις. Δεν έχουμε πια χρόνο. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, προστασίας, επεξεργασίας δεδομένων ε, και χρειαζόμαστε να ρυθμίσουμε και όλα τα θέματα τα συναφή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε να διευθετήσουμε και την προστασία δεδομένων στο θεσμικό πλαίσιο. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε την ε, συνεργασία των αστυνομικών αρχών μέσα στην Ευρώπη. Ε, αλλά εδώ έχουμε καταντήσει να είμαστε άγρια δύση. Ο ένας ε, ακολουθεί τις α διατάξεις, ο άλλος τις β, άλλους νόμους, άλλες εφαρμογές ε, μα δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται ο κανονισμός, χρειάζεται η οδηγία και πρέπει με αυτό το χρόνο να τακτοποιήσουμε αυτή την υπόθεση για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Ο πρόεδρος, Γιώσεφ, θα έχει τελευταίο το λόγο, ο Φερνάντο. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα είμαι σύντομος. Το πρώτο μου σχόλιο ουσιαστικά είναι ε, να δείξω ότι υπάρχει συνέχεια στην προσήλωση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και πακέτο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι και για τα νέα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δηλαδή να καταλάβουν ότι εμείς έχουμε εργαστεί για χρόνια ολόκληρα στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου για αυτό το θέμα και για ε, πολύ βάσιμους λόγους. Είχαμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη Συνθήκη της Λισαβόνας και λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει επιτέλους ένα πραγματικά νομοθετικό σώμα με νομοθετική εξουσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Μιλάμε πλέον σοβαρά για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το δεύτερο είναι όχι μόνο να δείξουμε τη συνέχεια αυτή τη δέσμευση και προσήλωση, αλλά να διευκρινίσουμε ότι έχουμε ξαναδεί ε, παρελκυστικές ε, τακτικές, ε, να καθυστερούν δηλαδή για χρόνια κάποιες καταστάσεις και να μην έχουμε πρόοδο. Λυπούμε πολύ, όπως έγινε με την οριζόντια διγέα για την ισότιμη μεταχείριση, την καταπολέμηση των διακρίσεων, που δεν έχει μέχρι σήμερα πάρει σάρκα και οστά. Το ίδιο ισχύει για τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Χρόνια ολόκληρα έχουμε θλιβερή καθυστέρηση και ολιγορία. Παρότι εμείς ε, ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, τονίσαμε το θέμα αυτό, δεν βλέπουμε στην άκρη του τούνελ φως. Για αυτό το πακέτο για την προστασία δεδομένων ε, δεν ξέρω γιατί θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει λόγο να καθυστερήσει το θέμα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία ολιγορούν, βάζουν εμπόδια, παρακολύουν την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Προσπαθούν να μπλοκάρουν την κοινή θέση. Ξεκινώντας από τη γενική προσέγγιση, αυτή τη συνολική προσέγγιση. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα θέματα που διακυβεύονται. Ο κανονισμός φαίνεται να είναι το μείζον. Η οδηγία όμως για τα κρατημέλη είναι ίσως το πιο σημαντικό. Καλό είναι λοιπόν που είμαστε πιο κοντά ε, στο να καταλάβουμε καλύτερα ε, ποια είναι τα σημαντικά ε, σημεία του κανονισμού, αλλά και με την οδηγία πρέπει επακριβώς να δούμε ποιους κόρτες δεσμούς πρέπει να λύσουμε ώστε να λειτουργήσει, να γίνει πράξη αυτό το πακέτο. Και Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά τις εργασίες του Συμβουλίου ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι τριμερείς διάλογοι. Πρώτος πράγματι καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία κρεμεί. Επόμενος. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήμουν υπουργό αρμόδιος για τα ζητήματα διοίκηση και ψηφιοποίηση. Εργάστηκα στην Πολωνία λοιπόν και για αυτήν την οδηγία και για αυτόν τον κανονισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι από τα σημαντικότερα έγγραφα που πρέπει να εκπονηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2013 και το σχετικό με τον προγραμματισμό των εργασιών του Συμβουλίου για την περίοδο 2014-2019 και γιατί λέγεται ότι το 2015 είναι η τελευταία διορία για, αυτή τη, για αυτό το πακέτο. Τώρα, στην κοινωνία τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη, συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ μήπως πριν ρυθμίσουμε τη μεταβίβαση δεδομένων δεν πρέπει να δούμε πρώτα την προστασία των δεδομένων. Γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινωνία. Αν θέλουμε επίση να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ω Ευρώπη στον τομέα τη επεξεργασία δεδομένων, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο σε πολλού τομεί, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία. για τη διασύνδεση επιχειρήσεων και προσδοκιών της κοινωνίας. Για το 2015 και το κατά πόσο θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει. Αυτό θα είναι μια λιδία λίθο για το πόσο καλά μπορεί να συνεργαστεί Κομισιόν, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Επομένω, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι κάτι το οποίο ε, είναι απολύτω απαραίτητο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λέει ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Προεδρίας εδώ ή μάλλον αποφεύγει να μας ε, ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, ότι μπορεί να παραταθεί, να επιμηκυνθεί, το δέχομαι, αλλά όχι να μην ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η δουλειά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, που ακούμε από ένα νέο μέλος ότι έχει πρακτική εμπειρία. Άννα, ήθελες να πεις το λόγο, αλλά Γιώζεφ θα είσαι τελικά στον κατάλογο. Γιώζεφ, είσαι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μάλλον δυσάρεστη. Συνέχεια μιλάμε για τις βέλτιστες πρακτικές και σίγουρα όλη αυτή η υπόθεση δεν είναι τέτοιο παράδειγμα. Κάθε άλλο από βέλτιστη πρακτική είναι και δείχνει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Εάν ε, δεν λειτουργούμε μαζί συνεργατικά δεν δουλεύει το σύστημα διαθεσμικά πρέπει να λειτουργούμε και με σεβασμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι εντυπωσιακό ότι η συζήτηση αυτή γίνεται και στους ε, οικονομικούς κύκλους. Έγινε μια μεγάλη έκθεση, η έκθεση του Ανοβέρου όπως ξέρετε και όλος τομέας ε, πιστεύει ότι επιγόντως χρειαζόμαστε ρύθμιση αυτών των προβλημάτων εδώ και χρόνια πιέζουν και λένε ότι επιτέλους ε, αντιμετωπίστε αυτό το θέμα. Επίσης εκπλήττουμε ότι σε άτυπες συζητήσεις με εκπροσώπους ή μέλη του Συμβουλίου ε, πολλές, ακούμε τη γνώμη ότι ε, δεν ξέρουν ε, πώς ε, να ρυθμίσουν αυτό το θέμα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτά είναι εντυπωσιακά πράγματα. Με εκπλήττουν ιδιαίτερα, διότι πολλοί από αυτούς έχουν και πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν τις δικές μας εργασίες ε, δίκαια και δεν αναφέρουν αυτά τα οποία έχουμε κάνει και τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και οι κύκλοι της βιομηχανίας, εμπορίου, οικονομική, όλοι και οι πολίτες ε, καίγονται, θέλουν να δουν να αυτά τα θέματα των δεδομένων το ταχύτερο και πιστεύουν ότι εδώ ε, παίζεται ένα παιχνίδι εις βάρος τους εδώ και χρόνια. Όλη αυτή η καθυστέρηση, ό, όλη αυτή η δισταγμή που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι είμαστε ανήμποροι και αδύναμοι και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε ζητήματα τα οποία μας καίνε. πολύ σύντομα, Άννα, γιατί έχουμε τους ομιλητές περιμένουν. Ακούστε, πιστεύω ότι πράγματι θα ήταν ενδιαφέρον αν οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη πλευρά η Αμερικανική πλευρά αν εκπληρωθούν. Γιατί αυτό θα δείξει εάν τέλο πάντων ε, συναντηθούν τα πνεύματα αυτά, που θα συναντηθούν. Πρέπει όμως να το δούμε πριν το πιστέψουμε. Και αν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση ε, ότι παναχωρεί το Συμβούλιο σε σχέση με αυτά που έχουν επιτευχθεί, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει αυτή η προθεσμία που ανέφερε ο συνάδελφος κύριος Μπόνι με το αμερικανικό ημερολόγιο. Δεν νομίζω ότι είναι θετικό ε, να καθυστερήσουμε. Εγώ δεν περιμένω και πολλές εξελίξεις. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα. Είναι προφανώς πολύ σημαντικό για την προστασία των πολιτών μας. και της νομοθεσίας μας. Αλλά και για τις ΕΠΑ έχει συνέπειες και πρέπει να εργαστούν περισσότερο, μόνο να συνεργαστούμε με τους ε, ομολόγους μας από το Κογκρέσο ή με την Αμερικανική ε, πλευρά, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, ε, τον ΙΠΑ, που θα μπορούσε να είναι σύμμαχός μας στο μέτωπο του αγώνα για την προστασία των, προσ... δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καταπολέμησης διαφόρων εισβολών. για να είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν θέματα από συναδέλφους αλλά και αυτό που είπε ο Τζόσεφ για τα κράτη-μέλη και τη στρατηγική για το μέλλον. Υπάρχει ένα αίσθημα ότι τώρα δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε απλώς το Συμβούλιο για το μεγαλύτερο νομοθετικό έργο του κομμάτι του Κοινοβουλίου. Πες μας τι κάνουμε ενώπιση του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Ευθύ εξ αρχή πρέπει να πω ότι για μας ευθύ εξ αρχή ήταν κάτι δεν ε, συμβαίνει απέναντι σε κάποια τρίτη χώρα. Συμβαίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίζουμε μόνοι μας ποιο θα είναι το νομοθετικό μας πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αναφέρθηκε η, εμπορική, η Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία, ε, είναι πρόσδεκτο και συμφωνούμε ότι ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανειλημμένως ανακοίνωσε ότι η προστασία των δεδομένων δεν θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε αυτό το πλαίσιο γιατί εμείς αναθεωρούμε το δικό μας πλαίσιο και θέτουμε κανόνες στην αγορά μας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας και ε, σκεφτόμενοι τα συμφέροντα των εταιριών μας, των οικονομιών μας, γιατί όπως επισημάνθηκε υπάρχει ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή απέναντι ε, μεταξύ των Ευρωπαίων και εταιριών από τρίτες χώρες που μπαίνουν στην εσωτερική αγορά και που εύκολα μπορεί να επιλέξουν μία από τις 28 δικαιοδοσίες, να βάλουν ένα, μια ταχυδρομική θηρίδα ή μια σύνδεση διαδικτυακή και να προσφέρουν υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κάναμε μια τόσο τόσο ευρεία συμφωνία που συνδύασε δύο πράγματα. Αφενό με την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι τα πρότυπά τους δεν θα κατέβουν αλλά θα ενισχυθούν και δεύτερον την ξεκάθαρη δέσμευση για ένα εναρμονισμένο, ενοποιημένο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα συνεχίσει και θα επικρατήσει μόνο αν συνεχίσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Και όπως το είπα ξεκάθαρα η συνένεση είναι απαραίτητη. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι και η προσέγγιση του Συμβουλίου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους είχαμε προβλήματα στο Συμβούλιο ή βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο ήταν επίσης ότι υπήρχαν θέματα που ετέθησαν τα οποία ήταν τελείως ε, ε, εκτός τόπου. Δηλαδή να μην ε, μόνο και μόνο για να μην ε, ακολουθήσουμε το δρόμο της ενοποίησης της ε, νομοθεσίας απλώς του, της διαίρεσής της. Ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό, αυτό, σε σχέση με αυτά που κάνει το Κοινοβούλιο και κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Το νόημα του άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που λέει ότι δεν υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς είτε τη συνένεση είτε κάποια νομική βάση που περιγράφει νόμιμο συμφέρον επεξεργασία, αλλά μας λέει ότι υπάρχουν ε, και εκτό αυτού τομεί επεξεργασία. Αυτό είναι τελείως έξω από τι κόκκινε γραμμές που έχει θέσει το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2011. Αν λοιπόν, καταλήξουμε, αν λοιπόν ε, ε, ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτές τις προτάσεις που είναι τελείως ε, εκτός του πεδίου συζήτησης δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο πολύ γρήγορα. Τέσσερα χρόνια για την οδηγία 95-46 αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι εκεί χρειάστηκε μια νέα διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο Αξελφός και άλλοι, έχουμε ανάγκη από το τριμερή διάλογο ακόμα. Και αν αναλάβει κανείς, αν, ε, αν επικρατήσει στο Συμβούλιο ε, η θέση του Κοινοβουλίου τα τέσσερα χρόνια είναι εντάξει, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είναι έτσι. Υπάρχει ανάγκη να ενωθούμε ναι. και αυτό θα γίνει αν ε, υπάρξει τριμερής διάλογος. Πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, επανειλημμένως είπαμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν τα ανοιχτά ζητήματα. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές παρεξηγήσεις ε, στην αρχή, όλοι το γνωρίζουμε και ο καθένας μας χρειάστηκε να μάθει ένα σωρό πράγματα γιατί το ζήτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο, εκατοντάδες άρθρα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία κανείς δεν μπορεί να είναι ε, σίγουρος ευθύς εξ αρχής, ότι τα γνωρίζει πολύ καλά. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι ουσιαστικό και αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα είναι μεγάλη μας χαρά. Ε, δεν νομίζω ότι η γραμματεία της Επιτροπής ε, μπορεί να έχει, θα έχει πρόβλημα αν ο πρόεδρος καλέσει έναν από τους υπουργούς που έχει κάποιο θέμα και που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου, με τα χαρά θα τους δεχτούμε και θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Εν τω μεταξύ, καθώς θα προχωρεί όμως τη δουλειά το Συμβούλιο, για να είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε. Χαίρομαι πολύ που η κυρία Λάουστιν θα είναι η εισηγήτρια της οδηγίας. Για μία ακόμα φορά θέλω να επαναλάβω ότι για μας είναι πακέτο. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν μαζί. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα ήταν αυθαίρετο να μη συμφωνήσουμε για ελάχιστα πρότυπα, τουλάχιστον στον τομέα της ε, δίωξης της επιβολής του νόμου εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Τάξη Ερευνών και αυτό που μπορούμε να δείξουμε είναι ότι το Κοινοβούλιο ήταν πρωτοπόρος στο να πιστεύει ότι θα υπάρξουν κοινά πρότυπα τα οποία θα ε, ε, εγκριθούν αργότερα για την προστασία των δεδομένων και αυτό το έκανε αναγνωρίζοντας ε, τα παραδεχόμενο θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση μέτρων έρευνα χωρί να τα γνωρίζει. Το Κοινοβούλιο έδειξε ότι θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία, ε, δείχνοντα εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη που θα θέσουν τα πρότυπα. Ω εκ τούτου προτείνω το ταχύτερο δυνατό μετά το καλοκαίρι να γίνει συνεδρίαση των σκιωδών για να δούμε πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές που δόθηκαν σήμερα και να προχωρήσουμε τον περισσότερο. Um, Ευχαριστώ Γιάν. Χρειάζεται κοινή στρατηγική για το πακέτο για την συνεργασία με τη γραμματεία της ομάδας. Πολλοί από τους σκιώδεις είναι σήμερα εδώ, τα ακούν αυτά, θα θέσουν το σημαντικό αυτό θέμα με σκοπό να επιστρέψουμε το σεπτεμβριο οκτωβριο και τότε θα γίνει και η συνεδρίαση των σκιωδών ε, ως, ε, ως ε, αντιπρόεδρος μπορεί να συμμετέ, πρέπει να συμμετέχει και στους συντονιστές. Οπότε θα, ε, το αναλάβεις και αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και όλους τους παρόντες που τήρησαν το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Και το επόμενο θέμα που συμφωνήσαμε με τους συντονιστές θα συζητηθεί και κλεισμένων θυρών. Τα νέα μέλη, αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν θέση συνέθεση πρέπει να αποχωρήσουν. Members and group staff. Sophie, don't give me a hard time. It's my first day. Έχουμε πέντε χρόνια μόνο ακόμα, λέει η κυρία Βέλτ. Θέλω να πω για τα πρακτικά ότι διαφωνώ θεμελιωδώς ότι το safe harbor αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί και κλεισμένων των θυρών πρέπει να έχουμε γραπτή δικαιολόγηση από την Κομισιόν, διότι αυτό συνάδει ασφαλώς με την ομολογία της διαφάνειας, γιατί θέλει και κλεισμένων των θυρών, γιατί εμπιστευτικά τα κείμενα κλπ. Αυτή τη στιγμή ούτε νομοθετούμε, ε, ε, απλώς συζητούμε. Το, ε, βρισκόμαστε λοιπόν σε πολύ άσκημη θέση και επισήμως ζητώ και να γραφτεί στα πρακτικά να μας δώσει η Κομισιόν γραπτή δικαιολογία. Ε, ο πρόεδρος λέει, έχω γραπτό σε τη δικαιολογία της Κομισιόν γιατί προέβλεπα μια τέτοια αντίδραση. Μα εάν είναι μια, ένα αντίγραφο της προηγούμενης δικαιολογίας, λέει είπε η κυρία Βέλ, δεν το θέλω, θέλω κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, για να σοβαρευτούμε, κάνουμε μία εξαίρεση για αυτή ειδικά τη συνεδρίαση και την κάνουμε και κλεισμένων των θυρών. Το Σεπτέμβριο όμως δεν θα είναι και κλεισμένο. Για αυτή τη συνεδρίαση ορισμένες πτυχές οι συντονιστές πίστεψαν ότι θα πρέπει να συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών, άλλες όχι. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι απόφαση των συντονιστών. Και ε, δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ε, του κεκλεισμένων ή όχι κεκλεισμένων των σειρών, ειδικά σε ένα θέμα όπως η όλη διαδικασία του Safe Harbor, το οποίο θέμα αυτό είναι και λίγο αμφιλεγόμενο. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την άποψή σας και γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για να ξέρουμε ακριβώς πότε και για ποιο λόγο θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Αυτές θα υπάρχουν από το Σεπτέμβριο και θα τις συζητήσουμε με την Κομισιόν. Η κυρία ε, Βέλτ. Ε, ναι, σας εμπιστεύομαι. Εντάξει, σήμερα είναι μία εξαίρεση, αλλά δεν πρόκειται εδώ, δεν είναι αρμοδιότητα των συντονιστών και το πώς αισθάνονται ε, εδώ ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη σημασία αυτού του θέματος. Αυτό είναι για τους πολίτες, ούτε για μένα ούτε για τον διπλανό μου. Εδώ πρόκειται για το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ξέρει τι γίνεται. Και εδώ ελπίζω να μας ακούνε. Να μας ακούτε. Εδώ λοιπόν αρνούμε στους συναδέλφους, το, τους πολίτες μας το δικαίωμα να παρακολουθούν και να ενημερωθούν για αυτό το καυτό θέμα ο πρόεδρος. Πρέπει να υπάρχει δικαιολόγηση. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος, ε, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, οι συντονιστές πήραν αυτή την απόφαση, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά ε, η, όλη η Επιτροπή θα συμμετάσχει στην επόμενη συζήτηση του θέματος αυτού το Σεπτέμβριο, που δεν θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ε, λοιπόν, όλοι η ιδέα αυτή τη προκαταρκτική συζήτηση ήταν να μην μπερδέψουμε τα νέα μέλη. Τώρα πιστεύω ότι του έχουμε κάτι.